εκφωνείται η ομιλία από έναν πρόεδρο της ε, Κομισιόν ο οποίος ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο αυτό μετά τις ε, ευρωεκλογές και θεωρώ πως ε, πραγματικά σπανίως είχαμε τόση αναμονή για αυτή την ομιλία και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για το ότι θα εκφωνήσει αυτή την ομιλία ένας πρόεδρος ο οποίος εξελέγει με μια νέα διαδικασία η οποία κατέστησε την Ένωσή μας πιο δημοκρατική. Το σώμα λοιπόν είναι και σήμερα το πρωί ο τόπος της ε, ευρωπαϊκής ε, δημοκρατίας και βεβαίως αντιμετωπίζουμε μια ιστορική πρόκληση για την αντιμετώπιση της κρίσης των ε, προσφύγων αλλά και της ε, οικονομικής κρίσης και θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τα κράτη με λύσεις. Η συζήτηση λοιπόν για την κατάσταση της ε, Ένωσης αφορά και την σχέση εργασίας μεταξύ Κομισιών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά επίσης είναι η στιγμή στην οποία τα δύο αυτά θεσμικά όργανα μπορούν να δείξουν ότι μπορούν να λειτουργήσουν με κοινοτικό πνεύμα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ σήμερα θα μας μιλήσει για πρώτη φορά με την ε, ιδιότητά του αυτή για την κατάσταση της Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, σας δίνω τον λόγο για να μας παρουσιάσετε τις προτάσεις που έχετε να κάνετε εσείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον οίκο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κυρίες μου και κύριοι βουλευτές, είναι ευχάριστο καθήκον, αλλά και ευχαρίστηση για μένα για πρώτη φορά ως πρόεδρος της Κομισιόν να εκφωνήσω αυτόν τον λόγο. Ως Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου πάρα πολύ συχνά, 20 φορές νομίζω, εκφώνησα λόγο για την κατάσταση του έθνους και πάντα μου λέγανε πως ήταν ε, πάρα πολύ, καλό, ε, πάρα πολύ καλός ο λόγος που εκφώνησα όσον αφορά την ρητορία και τον τόνο. Για το περιεχόμενο βεβαίως οι απόψεις ε, ήταν πάντα διαφορετικές και πάντα μου έλεγαν ότι μακρηγορούσα. Το ίδιο αναμένω να συμβεί και σήμερα. Για λόγους που φαντάζεστε Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένος. Κοιτάξτε, η ομιλία αυτή λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του τρόπου λειτουργία που έχει καθορίσει η διοργανική συμφωνία μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου και ορίζει ότι στο πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου θα πρέπει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λογοδοτήσει για τα όσα έχει κάνει μέχρι στιγμής και για τα όσα προγραμματίζει να κάνει τους επόμενους μήνες. Μιλάμε δηλαδή για τις ε, προτεραιότητες, για τις μελλοντικές εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άρα εν μέρη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για τον ε, σκοπό αυτό Έχω δώσει γραπτός ε, στον Μάρτιν Σούλτς ε, και στον ε, πρόεδρο της Λουξεμβουργικής Προεδρίας γραπτός τις προτεραιότητες μας. Και η επιστολή αυτή συνοδεύεται και μία παρουσίαση των δέκα προτεραιοτήτων της εργασίας της Κομισιόν. Λοιπόν, όλα αυτά δεν θα τα αναπτύξω σήμερα και σας παραπέμπω, μπορεί να μην είναι πάρα πολύ ευγενικό αλλά είναι αναγκαίο στην αλληλογραφία ε, μας στις επιστολές ε, τις οποίες ε, υπογράφω εγώ και ο αντιπρόεδρος ο κύριος Φρανς Τίμερμανς για να γίνει πιο κατανοητή η κατάσταση. Είμαι λοιπόν ο πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος διαζώσεις ε, και όχι με έμεσο αλλά με άμεσο τρόπο εξελέγηνα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 ε, ε, Ιουλίου πέρσι όταν και ξεκαθάρισα ότι η δική μου Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι πιο πολιτική και άρα ο πρόεδρος αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω του πιο δημοκρατικού τρόπου εκλογής του θα είναι και πιο πολιτικός πρόεδρος. Όταν λέω πολιτικός Το εννοώ με την ε, ευγενή έννοια της λέξης. Είμαστε πολιτικοί άνδρες και γυναίκες και δεν είμαστε πολιτικάντιδες. Και εσείς και εμείς είμαστε άνθρωποι που ασχολούμεθα με την πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι θα πολιτικοποιήσουμε τα πάντα. Αλλά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 εκφωνώ τη λέξη κοινωνικός να μην μετράτε πόσες φορές θα πω την λέξη αηφόρος, πόσες φορές θα πω την λέξη οικονομικός, χρηματοοικονομικός ή προϋπολογισμός. Συχνά ακούμε μεγάλα και κενά λόγια, αλλά πλέον νομίζω πως έχει φτάσει η ώρα της ειλικρίνειας στην Ευρώπη. Γι' αυτό θεωρώ πως ε, θα πρέπει να μιλήσω για τα μεγάλα, ανοιχτά, τεράστια ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτά θα επικεντρωθώ. Η Ευρωπαϊκή μας Ένωση, παρά το ότι δεν είμαι απεσιόδοξος, δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Δεν έχει νόημα ο πρόεδρος της ε, Κομισιόν ε, να μην είναι ειλικρινής απέναντι στους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών λαών και άρα της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Η Ένωση λοιπόν δεν είναι σε καλή κατάσταση. Χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζεται περισσότερη Ένωση σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει τώρα και να το κάνουμε εμείς από κοινού. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να τηρήσετε την εντολή που έχετε λάβει από τους Ευρωπαίους ε, ψηφοφόρους και να τιμήσουμε και εμείς την εντολή που λάβαμε από το σώμα. Μάλιστα. Μα δεν... δεν ξέρω γιατί εκνευρίζεστε όταν λέω τέτοια για περισσότερη ένωση. Α, καλά, καλά, καλά. Μπορείτε μερικές φορές να με διακόπτετε, αλλά δεν θα απαντάω συστηματικά σε αυτά που λέτε, γιατί αυτά που λέτε είναι ανάξια λόγου. Κύριε, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ό,τι προγράμματα εργασίας θα μπορούσαμε να καταστρώσουμε, η πρώτη προτεραιότητα σήμερα είναι το θέμα των προσφύγων. Από τις αρχές του έτους 500.000 περίπου άνθρωποι έφτασαν στην Ευρώπη from Syria. Οι περισσότεροι έφυγαν από τη Συρία, από την τρομοκρατία των δικτατοριών και την Ερυθρέα και τη Λιβύη. Πάνω από 200.000 έφτασαν από την Ελλάδα, την Ιταλία και μέσω Ουγγαρίας. Η αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Για μερικούς είναι και τρομερή, εκφοβιστική. Δεν είναι όμως τώρα ώρα και καιρός να φοβηθούμε, αλλά να δράσουμε συντονισμένα ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως κράτη-μέλη και ως θεσμοί. <clears throat> Το πρώτο θέμα, το κυριότερο, είναι θέμα ανθρωπισμού <clears throat> και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. <clears throat> Και για την Ευρώπη είναι και θέμα ιστορικής δικαιοσύνης. Εμείς οι Ευρωπαίοι, γιατί εδώ όλοι οι Ευρωπαίοι είμαστε, <laughs> ναι, ναι, καλά, καλά. Σημειώνω ότι εσείς δεν θεωρείτε τον εαυτό σας Ευρωπαίο. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι λοιπόν τώρα ο καιρός να φοβηθούμε. Αλλά να επιδείξουμε ανθρωπισμό και να καταλάβουμε την αξιοπρέπεια που πρέπει να αναγνωρίσουμε στις πρόσφυγες. Πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι η Ευρώπη είναι ήπειρος και όλοι σχεδόν οι κατοικοί της κάποια εποχή υπήρξαν πρόσφυγες. Η κοινή μας ιστορία έχει σημειώσει πολλές προσφυγικές καταστάσεις από Ευρωπαίους που ήθελαν να διαφύγουν από καταπίεση από τη Γαλλία ας πούμε τον 17ο αιώνα Εβραίους, Ρωμά Προτεστάντες και φυσικά τις δεκαετίες του 30 και 40 του περασμένου αιώνα. Οι Ισπανοί δημοκράτες που έφευγαν από την Ισπανία στη, στο νότο της Γαλλίας στα τέλη της δεκαετίας του 30 μετά την ήττα τους στον εμφύλιο. Ούγγροι επαναστάτες που έφευγαν στην Αυστρία και αλλού. Παντού, παντού στην Ευρώπη. μετά την εξέγερση κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος που και την ρωσική παρέμβαση με τα τάγκς. Τσέχοι, Σλοβάκοι που ήθελαν να φύγουν σε άλλες χώρες και στη δική μου μετά την καταπίεση της άνοιξης της Πράγας το 1968. Εκατεντάδες χιλιάδων αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους μετά και κατά τη διάρκεια των Ιουγκοσλαβικών πολέμων προς το τέλος του προηγούμενου αιώνα, όχι εκατοντάδες χρόνια πριν, αλλά στο τέλος του προηγούμενου αιώνα, την τελευταία του δεκαετία. Αυτά τα ξεχάσαμε, ότι υπήρχαν λόγοι για τους οποίους ζουν περισσότεροι άνθρωποι με το όνομα Μακδόναλντ στις Ηνωμένε Πολιτείε από ό,τι στην ίδια τη Σκοτία. Υπάρχει λόγος για τον αριθμό των Ονίλ και Μάρφη που ζουν εκεί αντί στην Ιρλανδία. Ξεχάσαμε ότι 20 εκατομμύρια Πολωνοί ζουν εκτός Πολωνίας επειδή υπέστησαν οικονομική καταπίεση και κατά τις ιστορικές αλλαγές που υπέφερε τόσο συχνά η Πολωνία. Ξεχάσαμε ότι μετά την καταστροφή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου 60 εκατομμύρια έγιναν πρόσφυγες μέσα στην Ευρώπη λόγω αυτής της τρομερής ευρωπαϊκής εμπειρίας. Η συνθήκη της Γενέβης ε, δημιουργήθηκε ακριβώς για να δοθεί άσυλο σε όσους πρόσφυγες αναγκαζόταν να φύγουν και να καταφύγουν εναντίον της καταπίεσης. Εμείς οι Ευρωπαίοι με αυτά και να γνωρίζουμε ότι η χορήγηση ασύλου σε πρόσφυγες είναι κάτι βασικό, ένα βασικό δικαίωμα από, τα βασικό, από τις βασικότερες διεθνείς και ευρωπαϊκές αξίες. Σας έχω ξαναπεί και εδώ και αλλού ότι πολύ σπάνια είμαστε περήφανοι για την ευρωπαϊκή μας κληρονομιά και το όραμά μας. Παρά τις αδυναμίες μας ή αυτός που θεωρούνται αδυναμίες σήμερα παγκοσμίω η Ευρώπη θεωρείται ως τόπος ασύλου. Η Ευρώπη σήμερα εκπροσωπεί την ελπίδα για μια πιο σταθερή ζωή από, για ανθρώπους που προέρχονται και από τη Μέση Ανατολή και από αλλού. Γι' αυτό μπορούμε να είμαστε περήφανοι και όχι να το φοβόμαστε. Η Ευρώπη σήμερα κυρίες και κύριοι παρά τις διαφορές που έχουν τα κράτη της είναι η πιο ευημερούσα και πιο σταθερή περιοχή του κόσμου. Όσοι επικρίνουν την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Οικοδόμηση, την Ένωση πρέπει να παραδεχτούν ότι είναι χώρος και τόπος ειρήνης και σταθερότητας και μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. γιατί έχουμε τρόπο να βοηθήσουμε όσους φεύγουν διωκόμενοι από πολέμους και καταπίεση. Θα πείτε βέβαια εντάξει αλλά η Ευρώπη δεν μπορεί να τους δεχτεί όλους. Πράγματι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί όλοι, όλα τα προβλήματα του κόσμου και να τα λύσει. Αλλά πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους προοπτική. Προφανώς είναι πρωτοφανής ο αριθμός των προσφύγων που έρχονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά είναι μόνο 0,11% του συνόλου του πληθυσμού της Ευρώπης. Στο Λίβανο, συγκριτικά, οι πρόσφυγες είναι το 25% των κατοίκων του αυτή τη στιγμή σε χώρα που έχει έκταση μόνο για την ευημερία του ενός πέμπτου της Ένωσης. Ποιοι νομίζουμε ότι είμαστε λοιπόν. Να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς προς τους πολίτες. Όσο υπάρχει πόλεμος στη Συρία και τρομοκρατία στη Λιβύη, η κρίση των προσφύγων θα συνεχίζεται. Μπορούμε να χτίσουμε τείχη και τείχους και σειρματοπλέγματα, αλλά φανταστείτε για λίγο, αν εσείς αναγκαζόσαστε να πάρετε το παιδί σας στα χέρια και να φύγετε, τι θα κάνατε θα πληρώνατε οποιαδήποτε, οποιοδήποτε τίμημα. Θα σκαρφαλώνατε όλους τους τοίχους και δεν θα σας εμπόδιζε καμία θάλασσα, κανένα σύνορο δεν θα διστάζατε να περάσετε. Γιατί εδώ πρόκειται για τη βαρβαρότητα του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους, παραδείγματος χάρη. Προσπαθούμε να το καταπολεμήσουμε, <clears throat> γιατί τότε να μην βοηθήσουμε και εκείνους που διαφεύγουν από τα νύχια του. Καιρός είναι να δράσουμε, να διαχειριστούμε την κρίση των προσφύγων, γιατί δεν έχουμε άλλη εναλλακτική. Λίγοι κατηγόρησαν. Αλλά λίγοι πρότειναν λύσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Χώρες μέλη αλληλοκατηγορήθηκαν ότι δεν κάνουν αρκετά ή ότι δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Δυστυχώς Κανείς βέβαια δεν τόλμησε να πει ότι οι Βρυξέλλες και οι Κομισιόν δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Θα μπορούσαμε σχεδόν όλοι, οι περισσότεροι και εγώ και η Επιτροπή μου, θα μπορούσαμε να θυμώσουμε για, αυτό, για αυτές τις κατηγορίες, αλλά τι νόημα θα είχε. Ο θυμός δεν βοηθάει κανέναν και η κατηγορία, οι αλληλοκατηγορίες επίσης δεν βοηθούν κανέναν. Συχνά αυτές οι κατηγορίες είναι τόσο πολλές που δεν αναγνωρίζουν καν ότι μπορεί οι πολιτικοί να έχουν ξαφνιαστεί από τις εξελίξεις. Υπάρχουν πράγματα που έχουν συμφωνηθεί και τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη σημερινή κατάσταση. Θα πρέπει να δούμε τι έχουμε στη διάθεσή μας και να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα. Δεν θα ξεκινήσουμε κάτι το καινούριο. Ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι η δική μου Επιτροπή αλλά η Επιτροπή του Μπαρόσο, επανειλημμένα έχει κάνει προτάσεις έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό σύστημα χορήγησης ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν τμηματικά σταδιακά υιοθετήσει για αυτές τις προτάσεις και το τελευταίο κομμάτι αυτής της διαδικασίας έγινε δεκτό και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2015, δύο μήνες δηλαδή έχουν περάσει από τότε. Έχουμε λοιπόν κοινά επίπεδα προβλέψει στο σύνολο της Ευρώπης. Για αυτούς που ζητούν άσυλο, σεβόμενοι την αξιοπρέπειά τους, και στις διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν. Και έχουμε κυρίως κοινά κριτήρια για να κριθεί αν κάποιος πράγματι μπορεί να τύχει εθνικής προστασίας, διεθνούς συγγνώμη προστασίας. Αλλά όλα αυτά τα επίπεδα προστασίας, τα κοινά, θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως και θα πρέπει να γίνουν σεβαστά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να καταστούν ευρωπαϊκή πρακτική. Αυτό σήμερα δεν ισχύει. Ή μάλλον πριν το καλοκαίρι δεν ίσχυε σε καμία περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ε, τις πρώτες από 32 ε, διαδικασίες επί παραβάση έτσι ώστε να πείσει τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει. Είναι θέμα αξιοπιστίας. Ε, αποφασίζουμε, νομοθετούμε και δεν εφαρμόζουμε. Είναι λοιπόν θέμα αξιοπιστίας και των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σεβαστούμε το κοινοτικό, το εθνικό και το διεθνές δίκαιο. Μια δεύτερη σειρά διαδικασιών επί θα ακολουθήσει σε λίγες μέρες. Το ότι έχουμε αυτά τα κοινά επίπεδα προστασίας είναι κάτι το αρκετά σημαντικό πράγμα, αλλά δεν φυσικά μας καλύπτουν στην παρούσα φάση της, προσ... της κρίσης των προσφύγων. Είχε πει το Συμβούλιο, η Επιτροπή μάλλον, την Άνοιξη ότι απαιτείται να υπάρξει μια κοινή ατζέντα για το ε, θέμα της μετανάστευσης. Κάναμε ε, κάποιες προτάσεις ε, τον Μάιο και από τότε θα ήταν άδικο να πει κάποιος ότι δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα. Νομίζω ότι έχουμε τριπλασιάσει την παρουσία μας ε, στις θαλάσσιες περιοχές. Έχουμε, χάσει, έχουμε ε, σώσει χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες από τότε. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούν να χάνονται ζωές, έστω και μία ζωή είναι μία παραπάνω από όσο πρέπει αλλά παρόλα αυτά έχουμε διασώσει πολύ περισσότερο κόσμο κατά 250% και δεν πρέπει να το κρύβουμε, πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τις επιδόσεις μας αυτές. Ε, πάρα πολλές κοινοτικέ χώρες ε, και του Σέγγεν και εκτός συμμετέχουν, ε, ξέρετε, στις προσπάθειες του Frontex υπάρχουν πάνω από 100 αξιωματικούς, 30 σκάφη, 4 ελικόπτερα και υπάρχουν επίσης και διάφορα αεροσκάφη μεταφορικά και παρακολούθησης τα οποία αποδεικνύουν θα έλεγα ότι υπάρχει αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα. Έχουμε επίσης ε, επιτεθεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στις ομάδες των εγκληματιών που εκμεταλλεύονται αυτούς τους ανθρώπους. Αυτά οδηγούν βέβαια στο να χρησιμοποιούνται όλο και πιο μικρά σκάφη ε, τον Αύγουστο είχαμε γύρω στις 150.000 αφήξεις, κάτι το οποίο είναι αντίστοιχο με τον προηγούμενο χρόνο, αυτά όμως για την Νότια Μεσόγειο. Το θέμα είναι να συμβεί το υπόλοιπο και στις υπόλοιπες περιοχές της Μεσογείου ε, και επίσης να δούμε τι θα κάνουμε και συνολικά με το θέμα των εξωτερικών συνόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη δωρήτρια δύναμη στον κόσμο για την βοήθεια της, των προσφύγων από την ε, Συρία. 4 δις ευρώ έχουν κινητοποιηθεί μέχρι σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή και από εσά και από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές βοήθειας ανθρωπιστικής και οικονομικής προς τους Σύρους, προς τους πρόσφυγες και στις γειτονικές χώρες όπως το Ιράκ, το Λίβανο, την Ιορδανία, την Τουρκία και την Αίγυπτο. Και σήμερα μάλιστα ξεκινήσαμε και δύο νέα προγράμματα ε, για τη σχολική εκπαίδευση 240.000 ε, παιδιών προσφύγων στην Τουρκία. Και εδώ θα ήθελα να χειροκροτήσω τις προσπάθειες τις οποίες κάνει η Ιορδανία, η Τουρκία ε, και οι υπόλοιπες όμορες χώρες Οι χώρες αυτές, οι οποίες είναι πολύ φτωχότερες από μας, παρόλα αυτά κάνουν τεράστιες προσπάθειες τις οποίες θα πρέπει να χειροκροτήσουμε και να αναγνωρίσουμε και σε επίπεδο δεοντολογίας και σε επίπεδο οικονομικό. Έχουμε λοιπόν εμείς αναλάβει την υποχρέωση να υποδεχθούμε 22.000 ε, άτομα τον επόμενο χρόνο από την περιοχή αυτή αποδεικνύοντας έμπρακτα τις μορφές αλληλεγγύης. Αυτό φυσικά ε, είναι πάρα πολύ μικρός αριθμός σε σχέση με τις τεράστιες προσπάθειες που κάνουν αυτές οι άλλες χώρες όπως η Τουρκία, η Ορδανία και ο Λίβανος που έχουν υποδεχθεί μέχρι τώρα 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Παρ' όλα αυτά όμως ξεκινάμε την διαδικασία και θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε ε, τις προσπάθειες επανεγκατάστασης των προσώπων αυτών. Αυτό θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε ένα διαρθρωμένο σύστημα ε, επανεγκατάστασης και ένα πιο συστηματικό τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακόμα πολλά περιθώρια επίδειξης αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες οι οποίοι έρχονται στις χώρες μας. Είναι σαφές για μένα ότι τα κράτη-μέλη ε, στα οποία φτάνουν πρώτα οι πρόσφυγες, δηλαδή η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ουγγαρία, δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθούν ε, για να αντιμετωπίσουν αυτήν την τεράστια πρόκληση. This is why the commission... Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει εδώ και αρκετούς μήνες ένα μηχανισμό κατεπήγοντος, κατεπήγοντα μηχανισμό λοιπόν για την υποδοχή 40.000 ανθρώπων που ζητούν διεθνή προστασία και που βρίσκονται στην Ελλάδα και την Ιταλία και γι' αυτό σήμερα προτείνουμε ένα δεύτερο κατεπήγοντα μηχανισμό για περαιτέρω 120.000 άτομα από την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία. Αυτό θα πρέπει να γίνει με δεσμευτικό τρόπο. Απευθύνομαι λοιπόν προς τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατεπίγουσα επανεγκατάσταση των 160.000 προσφύγων συνολικά στη συνάντησή τους την 14η Σεπτεμβρίου. 120 ε, συν 40 μας δίνει 160.000 θα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους αυτούς θα πρέπει να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους αυτούς και ελπίζω σε αυτή την περίπτωση όλοι να πάρουν μέρος στην προσπάθεια. Να μην υπάρξουν απομονωτικές ρητορικέ. Αυτό το οποίο απαιτείται είναι δράση. What is happening to um, human beings? We are talking τι συμβαίνει στους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει. Δεν μιλάμε για αριθμούς, μιλάμε για ανθρώπους. Αυτοί που έρχονται από τη Συρία είναι άνθρωποι. Και αυτό θα μπορούσε να συμβεί αύριο σε άλλες περιοχές, στην Ουκρανία σαν παράδειγμα. Δεν μπορούμε να είμαστε επιλεκτικοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις ανάμεσα σε Ισραηλίτες, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους. Εμείς έχουμε θέσει τέλος στις θρησκευτικέ διακρίσεις. Δεν λαμβάνουμε σε σχέση με τους πρόσφυγες υπόψη μας τη φιλοσοφία του καθενός ή την θρησκεία του καθενός. Κυρίες και κύριοι, πλησιάζει ο χειμώνας όμως. Θέλουμε να υπάρχουν ε, τον χειμώνα οικογένειες να κοιμούνται σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε κρύες ε, σκηνές. Ε, θέλουμε είτε στη Βουδαπέστη είτε στο, στην Κο είτε σε άλλα μέρη. Πρέπει λοιπόν να προλάβουμε τη χειμερινή περίοδο και να φροντίσουμε αυτούς που φεύγουν από την καταστροφή που χτυπάει τις χώρες τους. Φυσικά το θέμα της επανεγκατάστασης δεν λύνει από μόνο του το πρόβλημα. Είναι επίσης ανάγκη είναι επίσης ανάγκη να βρούμε ένα ευρύτερο σύστημα προστασίας αυτών που εγκαταλείπουν τις χώρες τους. Ακόμα και ε, και αυτούς οι οποίοι φεύγουν από τις χώρες τους για λόγους που δεν τους δίνουν την δυνατότητα να ζητήσουν άσυλο. Και γι' αυτό προσέχουμε ακριβώς να φτιάξουμε τον κατάλογο αυτό των χωρών προέλευσης. αυτό θα περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία θα μας δείχνουν ποιες είναι οι χώρες οι οποίες υποτίθεται παρέχουν ασφαλείς τρόπους ε, επιβίωσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο ίδιος κατάλογος και τα ίδια κριτήρια της Κοπενχάγης στη συγκεκριμένη περίπτωση από όλες τις χώρες και σε επίπεδο δημοκρατίας και σε επίπεδο κράτους δικαίου και σε επίπεδο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. να λάβουμε υπόψη μας και την πρόοδο σαν παράδειγμα η οποία έχει υπάρξει σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων τα τελευταία χρόνια. Ο κατάλογος των ασφαλών αυτών χωρών λοιπόν είναι μια διαδικαστική θα έλεγα απλούστευση ε, του τρόπου με τον οποίο κρίνουμε το δικαίωμα χορήγησης ασύλου ανθρώπων που προέρχονται από τη Βοσνία Ερσεγοβίνη, από την Αλβανία, από την τέως Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, από το Κωστικοπαίδιο, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την Τουρκία. Αλλά παρόλα αυτά θα επιτρέψει στις εθνικές αρχές αυτή η λίστα στην παρούσα φάση να αντιμετωπίσουν με ενιαίο τρόπο αυτούς τους ανθρώπους σε σχέση με αυτούς οι οποίοι προέρχονται από χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση όπως τη Συρία. Ο κατάλογος ε, των ασφάλων χωρών οπωσδήποτε δεν αφαιρεί δικαιώματα του ασύλου από τις χώρες που περιέχονται σε αυτό τον κατάλογο. Είναι σημαντικό αυτό. Το άσυλο είναι δικαίωμα. Δεν υποσκάπτουμε τη συνθήκη της Γενέβης. Και οι χώρες που θα είναι στον κατάλογο αυτών πρέπει να γνωρίζουν πως εάν βγουν από αυτόν τον κατάλογο επειδή παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα παραδείγματο χάρη χάνουν την ευκαιρία να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά πάνε μαζί. Ασφαλής χώρα, ναι. Αλλά έχει φτάσει η στιγμή να γίνει μια πιο θεμελιώδης ε, αλλαγή στο πώς ε, κρίνουμε τις αιτήσει ε, ασύλου και συγκεκριμένα το σύστημα του Δουβλίνου που λέει πως τις αιτήσει πρέπει να τις κρίνει η πρώτη χώρα εισόδου. Χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη στην πολιτική ασύλου, περισσότερη ένωση στην πολιτική προσφύγων. Εδώ λοιπόν απαιτείται άλλη λεγγύη σε μόνιμη βάση και στους κανόνες και στην πολιτική μας. Γι' αυτό σήμερα η Κομισιόν επίσης προτείνει έναν μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης ο οποίος θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίζουμε κρίσεις πιο γρήγορα στο μέλλον. Πιο γρήγορα, ενώ πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν. Μια κοινή πολιτική προσφύγων και ασύλου, σημαίνει περαιτέρω προσέγγιση των ε, πολιτικών αφού αποδοθεί το καθεστώς του πρόσφυγα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να ξαναδούν τους μηχανισμούς στήριξης και ένταξης. Η Κομισιόν είναι έτοιμη να εξετάσει το πώς ε, θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτούς τους στόχους. Και είμαι υπέρ, υπέρ του να επιτρέψουμε στους ετούντες άσυλο να εργαστούν, να εργάζονται ενώ όσο περιμένουν να ακριθεί η αίτησή τους. Work. Η εργασία, η δουλειά είναι θέμα αξιοπρέπειας. Όσοι δουλεύουν ξαναβρίσκουν την αξιοπρέπειά τους. Οπότε πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να αλλάξουμε την εθνική νομοθεσία για να επιτρέψουμε, να, επιτρέψουμε στους ε, πρόσφυγες να δουλεύουν. Μια ενιαία πολιτική προσφύγων και ασύλου επίσης απαιτεί εντονότερες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Ευτυχώς εντός της Ένωσης δεν υπάρχουν ε, συνοριακή έλεγχη στην ζώνη Σέγγεν για να εγγυόμαστε ακριβώς την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών και το σύστημα Σέγγεν δεν θα καταργηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας της δικής μου επιτροπής. Αλλά η άλλη όψη του νομίσματος της ε, ελεύθερης ε, μετακίνησης είναι πως θα πρέπει να συνεργαστούμε στενότερα για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Αυτό περιμένουν από μας οι πολίτες μας. Εγώ το είπα στην προεκλογική εκστρατεία μαζί με τον Μάρτιν, τον Γκί και... Όχι. Δεν δείχνω την κυρία Κέλλερ. Ε, έψαχνα τον κύριο Τσίπρα σκεφτόμουν. Δεν, δεν τους μπερδεύω, μη φοβάστε. Ορίστε. Ναι, ο Ζωζέ Μποβέ είναι εδώ. Ναι, ναι, τον είδα, τον είδα. Συγγνώμη, Ζωζέ. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε πολύ τη Frontex και να γίνει μια πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή συνοριακή φύλαξη και ακτοφυλακή. Αυτό είναι εφικτό, αλλά βεβαίω σημαίνει πως χρειάζονται λεφτά. Η Κομισιόν θεωρεί πως είναι μια καλή επένδυση και προτείνουμε φιλόδοξα βήματα για μια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή και συνορία και θα τα προτείνει πριν το τέλος του έτους. Επίσης, μια ενιαία πολιτική μετανάστευση σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα διανοίξουμε νόμιμες διόδους. Αλλά ας είμαστε σαφείς. Αυτό δεν θα βοηθήσει την αντιμετώπιση, στην αντιμετώπιση της κρίσης των προσφύγων. αλλά εάν έχουμε ασφαλείς διόδους προς την Ευρώπη θα διαχειριστούμε καλύτερα τις ροές και θα καταστήσουμε λιγότερο ελκυστικούς τους διακινητές. Μην ξεχνάμε πως πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση της ε, δημογραφικής φτύσης. Χρειαζόμαστε ταλέντα από όλο τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν η μετανάστευση να αλλάξει από ένα πρόβλημα που χρειάζεται αντιμετώπιση προς έναν πόρο προς διαχείριση. Για το σκοπό αυτό η Κομισιόν θα προτείνει ένα πακέτο νόμιμης μετανάστευσης το 2016. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Κομισιόν θα πρέπει να νομοποιηθεί. Δεν έχει νόημα να παραπονιόμαστε για την παράνομη μετανάστευση. Πρέπει να οργανώσουμε και την νόμιμη μετανάστευση. A lasting solution will only come Μια διαρκής λύση θα επέλθει μόνο όταν αντιμετωπίσουμε τις αιτίε. Γιατί αντιμετωπίζουμε αυτή την κρίση, την προσφυγική. Πρέπει λοιπόν η ευρωπαϊκή πολιτική να είναι πιο στιβαρή, η εξωτερική πολιτική να είναι πιο στιβαρή. Δεν μπορούμε πλέον να αγνοούμε τους πολέμους και την ε, αστάθεια στη γειτονιά μας. Πρέπει να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα της Λιβύης. Δεν ξέρω, ίσως να είμαστε πάρα πολύ αδύναμοι για να κάνουμε κάτι. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την κρίση της Συρίας πιο αντέτικα. Θα πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική επίθεση για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στη Λιβύη και στη Συρία. Χρειαζόμαστε μια πιο ισχυρή Ευρώπη λοιπόν στην εξωτερική πολιτική. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι η Φεντερίκα Μογκερίνη, η ύπατη εκπρόσωπος, την έχει προετοιμάσει το έδαφος για μια τέτοια πρωτοβουλία. και επίσης είχε μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία όσον αφορά τις ε, συνομιλίες ε, για το Ιράν και θα ήθελα εδώ πέρα να την ε, συγχαρώ γι' αυτό. Για να διευκολύνουμε λοιπόν το έργο της είπα της εκπροσώπου μας, ε, της ε, Φεντερίκα, η Κομισιόν σήμερα προτείνει να συσταθεί ένα ταμείο ανάγκης με αρχικό κεφάλαιο 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για να αντιμετωπίσουμε την κρίση στο Σαχέλ, στο κέρας της Αφρικής, στην περιοχή των μεγάλων λιμνών της Αφρικής, για να δημιουργήσουμε σταθερότητα μέσω παραδείγματος χάρη ε, της ε, απασχόλησης στις τοπικές κοινότητες και άρα να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες της αστάθειας ε, των εκτοπισμών και της παράνομης μετανάστευσης. Και αναμένω από όλα, όλα τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν σε αυτό το ταμείο. Χρειαζόμαστε αυτό το ταμείο για να προλάβουμε μελλοντικές κρίσεις. And we Και χρειαζόμαστε επίσης περισσότερη ανάπτυξη και αναπτυξιακή βοήθεια. Δεν μ' αρέσει η έκφραση, αλλά προϋπολογισμούς συνεργασίας, ας πούμε. Δεν είναι φυσικό να μειώνονται οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών όσον αφορά την ανάπτυξη. Πρέπει να αυξηθούν. Δεν θέλω κύριε Πρόεδρε να δημιουργήσω αυταπάτες ότι η κρίση των προσφύγων θα τελειώσει σύντομα. Δεν θα τελειώσει σύντομα και πρέπει να το ξέρουμε αυτό αλλά να και με καταβλισμούς προσφύγων να διώχνουμε πλοιάρια, αυτό δεν είναι Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ο φουρνάρης στην κόπο που έδωσε δωρεάν ψωμιά στους πρόσφυγες. Είναι οι φοιτητές στο Μόναχο και στο Πάσαο που υποδέχτηκαν στο σταθμό τους πρόσφυγες. Αυτό είναι η Ευρώπη, εκείνοι που περίμεναν στο σταθμό του μονάχου χειροκροτώντας <coughs> την αύξηση των προσφύγων. σε αυτή την Ευρώπη εγώ θέλω να ζήσω που δείχνουν αυτά τα παραδείγματα και η Ευρώπη στην οποία δεν θέλω να ζήσω είναι μια Ευρώπη που αρνείται πρόσβαση σε κόσμο που έχει ανάγκη. Φυσικά θα διαρκέσει ακόμα η κρίση αυτή και υπολογίζω και σε εσά εδώ μέσα στο ναό αυτό της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας για να συνεργαστείτε κι εσείς με την εφαρμογή των κοινών μας στόχων. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτέ ή και αγαπητοί φίλοι για ορισμένους. Συνήθως όταν μιλάει ο πρόεδρος της Κομισιόν για την κατάσταση της Ένωσης του δίνουν λιγότερο χρόνο αλλά επειδή η κατάσταση είναι σοβαρή χρειάστηκα παραπάνω. Και η συζήτηση που έχει γίνει πολλές φορές λόγω, να προσθέσω ένα θέμα ακόμα, το, του ελληνικού προβλήματος ήταν πολύ δύσκολη διότι συνεχώς προσπαθούσα να εξηγήσω στον τότε Πρωθυπουργό ότι στην Ευρωζώνη υπάρχουν 19 δημοκρατίες και όχι μόνο η ελληνική οι διάφορες κοινέ γνώμες και οι βουλές εκφράζονται και από τις 18 άλλες χώρες που ανήκουν στην Ευρωζώνη. Συχνά η Κομισιόν έχει τύχει επιθέσεων από ορισμένε χώρες μέλη για τον τρόπο με τον οποίο πλάκι στην λύση, αν και δεν υπάρχει ακόμα λύση, του ελληνικού προβλήματος. Θέλω να επαναλάβω λοιπόν και το λέω και ενώπιόν σας, το είπα και όταν ήρθα την πρώτη φορά να σας μιλήσω, ότι καθήκον της Κομισιόν είναι να φροντίζει το γενικό συμφέρον. Να μην ασχολείται να μην ασχοληθούμε με το ελληνικό πρόβλημα θα ήταν απαράδεκτο λάθος και αδυναμία αν δεν είχαμε κάνει ό,τι κάναμε. Πληρώσαμε και εγώ προσωπικά ένα τίμημα αρκετά βαρύ αλλά όσον αφορά τις προσπάθειές μας αλλά δεν ήθελα να τα αφήσω όλα στα χέρια των ε, γραφειοκρατών των Βρυξελών αν και χρειάστηκε πάρα πολλή δουλειά ακόμη και κατά τις διακοπές δεν ήθελα μόνον οι γραφειοκράτες να ασχοληθούν με το πρόβλημα αυτό με τη λύση του ελληνικού προβλήματος επομένως και ο Τίμερμαν σε και ο Ντομπρόσκης και ο Πιέρ Μοσκοβισή και εγώ και άλλοι κάναμε πολλά για την επίλυση του ελληνικού προβλήματος που είχαμε μπροστά μας. Το να λέει κανείς ότι η Κομισιόν και ο Πρόεδρος της θεωρούν ότι το Brexit δεν είναι επιλογή μπορεί μεν να γίνει αλλά για μας δεν είναι επιλογή. Αλλιώς θα είχε γίνει ήδη. Και είπα στον κύριο Τσίπρα και στις ελληνικές αρχές ότι δεν πρέπει να θεωρήσουν τη φράση αυτή σαν να εννοεί ότι ούτως ή άλλως θα διασωθεί. Είπα στον Αλέξη Τσίπρα ότι εγώ δεν είμαι μάγος και ταχυδακτηλουργός που βγάζει λαγούς από το καπέλο του. Όχι. Ήξερε ότι το Brexit ήταν μια πιθανότητα αλλά που δεν θα αναφερόταν δημόσια. Και επ' αυτού κάναμε ό,τι έπρεπε και θεωρώ ότι το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι μόνο θέμα εξυγίανσης των δημοσιονομικών της χώρας, δεν είναι μόνο δομικό, αν και είναι σοβαρά όλα αυτά, αλλά είναι και πρόβλημα που αφορά τις δυνατότητες οπτικές ανάπτυξης της χώρας και θα έπρεπε η Ένωση να θεωρεί ότι έγινε ότι έπρεπε. Δεν μου άρεσαν τα σχόλια που έλεγα δεν έχει Ελλάδα παρά να βγει από το ευρώ σαν να μην είναι σοβαρή χώρα. Οι Έλληνες και μάλιστα κυρίως των χαμηλών εισοδημάτων εργάζονται σκληρά και κάνουν ό,τι μπορούν για να προοδεύσει η χώρα τους. Πρέπει λοιπόν να τους σεβόμαστε περισσότερο. Θα ήθελα το πρόγραμμα που συμφωνήσαμε να γίνει σεβαστό από οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο την προηγούμενη, όχι μόνο την τωρινή και όχι μόνο την επόμενη, όλες. Εάν αυτή τη φορά οι κοινοί κανόνες δεν γίνουν σεβαστοί, τότε η αντίδραση της Ένωσης και της Ευρωζώνης θα είναι διαφορετική. Αυτή τη φορά πρέπει να γίνει αυτό που συμφωνήθηκε. Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχουν 35 δισεκατομμύρια που οργανώνει η Κομισιόν για την αναθέρμανση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της ελληνικής δημοκρατίας. Και θα ήθελα η προσφορά αυτή, που δεν είναι βέβαια πλήρως δωρεά, να γίνει αποδεκτή από όλους τους ενδιαφερόμενους στην Ελλάδα. Η κρίση βέβαια δεν έχει τελειώσει με τη συμφωνία. Εφόσον υπάρχουν ακόμη 23 εκατομμύρια Ευρωπαίων που είναι άνεργοι και 17 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, στην Ευρωζώνη που δεν έχουν δουλειά, δεν τέλειωσε η κρίση. Θα τελειώσει την ημέρα που η Ευρώπη θα έχει επανέλθει στην πλήρη απασχόληση. Καμιά φορά αναρωτιέμαι πώς μπορεί μια τόσο πλούσια ήπειρο σαν την Ευρώπη να απομακρύνεται από αυτόν τον κανόνα που θα έπρεπε να γίνεται σεβαστό παρτού ότι οι νέοι και οι υπόλοιποι έχουν δικαίωμα στην πλήρη απασχόληση. Ας μην ξεχάσουμε αυτή την πρόθεσή μας να γίνει η Ευρώπη μία Ήπειρος όπου το τριπλό κοινωνικό α θα εφαρμόζεται παντού. Δεν είναι αδύνατο να επανέλθει η Ευρώπη στην πλήρη απασχόληση, αν το θέλουμε όλοι. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι θα παραμείνουμε πιστοί στην δημοσιονομική εξυγίανση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στις επενδύσεις. Έχουμε προτείνει και σε εσά και στο Συμβούλιο ένα επενδυτικό σχέδιο που αφορά 315 δισεκατομμύρια και το οποίο έχει αρχίσει να εφαρμόζεται γενικά και όσοι οι, όλοι οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών και οι επιχειρηματίες πρέπει να μπουν στη μάχη στον αγώνα για την ανάπτυξη της Ευρώπης. Το επενδυτικό σχέδιο που διεστυχώς φέρει το όνομά μου το λένε σχέδιο Juncker. Γιατί, για να βρουν έναν υπεύθυνο από διοπομπαίο τράγο αν αποτύχει. Θα ήθελα όμως όλοι οι οικονομικοί παράγοντες να εμπλακούν σε αυτό το επενδυτικό σχέδιο που είναι για την Ευρώπη και για την ανάπτυξη και για την απασχόληση. Όλα αυτά βέβαια κυρίε και κύριοι βουλευτές δεν αρκούν. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ορίσουμε, να χαράξουμε τον δρόμο τον οποίο θα ακολουθήσουμε στο μέλλον. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο προτείναμε το πρόγραμμα των λεγόμενων πέντε προέδρων για την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής και Οικονομικής Ένωσης. Αυτό το είπαμε πέντε προέδρων για λόγους αρχής. Ότι και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε προσωπικό επίπεδο θα πρέπει να εμπλακεί στην σύνταξη της συγκεκριμένης έκθεσης. Το κοινοβούλιο είναι ένα κοινοβούλιο και το να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να υπάρξει μέλλον στην Ευρώπη και μπορεί να υπάρξει εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την άμεση εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήταν εντελώς λάθος. Και γι' αυτό λοιπόν ενέπλεξα τον κύριο Σούλτς στις ε, εργασίες μας, ε, εξέφασε τις απόψεις του, δεν μου άρεσαν όλες, αλλά παρόλα αυτά έβαλε στη συζήτηση τη διοργανική τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν επανειλημμένα εκφραστεί από σας όπως τις απόψεις του κυρίου Ότμαρ Κάρας, σύμφωνα με την έκθεση που έγινε δεκτή στο όνομά του. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην χάραξη του ευρωπαϊκού μέλλοντος θα είναι σημαντική. Απαιτείται μια οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Δεν το λέω για πρώτη φορά, το λέω από το 1991 αυτό, από τότε που ήμουν Υπουργό Οικονομικών της χώρας μου με τον Νίκολα Σμιτ, ο οποίος ελέγχει τα πάντα στη χώρα μου εδώ και δεκαετίες. Ήμουν υπεύθυνο ε, για τη διακυβερνητική διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε και τέσσερις είχαν πει υπέρ. Ο Ζακ Ντελόρ, που είναι πάντα το πρότυπό μας, ο Πιέρ Μπερεγκοβουά, του οποίου η εξαφάνιση μας πείραξε όλους, ο Φιλίπ Μεστάτ, που είναι πάντα εδώ και μπορεί να μας διαφωτίζει με την πείρα του. Και εγώ ήμουν ο τέταρτος ακόμα εδώ. Είμαι συνεχώς παρόν αυτό. Το βλέπετε. Εν πάση περιπτώσει εμείς οι τέσσερις θέλαμε να εγγράψουμε στις συνθήκες κάποιους κανόνες οι οποίοι θα έπρεπε να χαρακτηρίσουν την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε δεν γίναν δεκτές οι απόψεις μας. τώρα έχουν αρχίσει να ε, συζητούν ε, για το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης διάφοροι. Ε, εντάξει, κάλιο αργά παρά ποτέ, το είχαμε πει πριν 25 χρόνια. Θα σας προτείνουμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα μέτρα για την ευάθυνση της Οικονομικής Ένωσης και ένα σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα, το κοινό σύστημα εγγύησης καταθέσεων, είναι απαραίτητο για το μέλλον μας. Θα το κάνουμε αυτό και είμαι βέβαιος με ένα σύστημα επανασφάλισης, όχι αμοιβεοποίησης, αλλά θα απαιτηθεί ένα επίπεδο επιπλέον ασφάλειας για τους καταθέτες στην Ευρώπη. Και θα το κάνουμε αυτό. Είμαι επίσης ε, υπέρ και ενός ε, λογιστηρίου ευρωπαϊκού θα έλεγα. Βέβαια είναι ένα σύνθημα στην παρούσα φάση αυτό το οποίο λέω. Δεν του έχουμε δώσει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο οικονομικό κέντρο αν θέλετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες σε καθημερινή βάση. Τώρα σε σχέση με τα δημοσιονομικά. όχι την δημοσιονομική πολιτική, αλλά τις δημοσιονομικές πολιτικές. Εδώ δεν υπάρχει ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταστήσει, σαν παράδειγμα στο θέμα το φορολογικό, το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις χώρες της Ένωσης να υιοθετηθεί το ταχύτερο δυνατόν από το Συμβούλιο. Εγώ εμένω σε αυτά τα οποία έλεγα και πίστευα όταν ήμουν 18 ετών. Κάποιοι πίστευαν ότι άλλαξα από τότε, δεν έχω αλλάξει. Τα κέρδη θα πρέπει να φορολογούνται στις χώρες στις οποίες παράγονται. Αυτή είναι η βασική αρχή και πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες. Θα πρέπει επίσης να αναλάβουμε δράση υπέρ ενός απλού κανόνος, ο οποίος απέδειξε ε, την ε, αποτελεσματικότητά του και την ωφέλειά του. Θα πρέπει δηλαδή στο σύνολο της Ευρώπης οι κανόνες αυτοί να γίνουν σεβαστοί. Ότι δηλαδή ίση εργασία στη συγκεκριμένη χώρα απαιτείται ίδια αμοιβή. Είναι παλιός ο κανόνας αυτός και θα πρέπει να εφαρμοστεί επιτέλους. υπό την καθεδήγηση και της κυρίας Τάισεν, της Επιτρόπου για Κοινωνικές Υποθέσεις. Εμείς θα προτείνουμε κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016 ένα ελάχιστο επίπεδο κοινωνικών δικαιωμάτων. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο το νόμισμα, δεν είναι μόνο η Ουκρανία, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα επίπεδο κοινό αξιών δικαιωμάτων που θα πρέπει να το καθιερώσουμε και να το υιοθετήσουμε. Έχω ένα πρόβλημα, Πρόεδρε. Σοβαρό πρόβλημα. Ξέρω, εσείς εκ δεξιών θα θέλατε να σταματήσω να μιλάω. Αλλά είμαι στη μέση της ομιλίας μου. Θα προσθέσω λοιπόν με μεγάλη ταχύτητα το εξής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παραμείνει το κοινοβούλιο της ζώνης ευρώ. Ας μην συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση με νέα στοιχεία κάνω μια απλή επιλογή αυτών που θέλω να σας πω. Γι' αυτό καθυστερώ. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο η διεθνής εκπροσώπηση της ζώνης ευρώ να βελτιωθεί από ό,τι σήμερα. Δεν είναι φυσιολογικό ε, στους θεσμούς του Bretton Woods και ιδιαίτερα στα πλαίσια του Δέλτα Νιτάφ η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρουσιάζεται με εντελώς ετερόκλητες απόψεις και κάθε χώρα τρέχει δεξιά-αριστερά όπου θέλει. Όχι, θα πρέπει ο πρόεδρος του Eurogroup να εκπροσωπεί μόνος του τη ζώνη ευρώ. Απαιτείται μια ενιαία μορφή εκπροσώπησης της ευρωζώνης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα πρέπει επίσης η αναχώραση στάσης τις οποίες αποφασίζει το Συμβούλιο και η Επιτροπή να γίνονται αντικείμενο καλύτερου σεβασμού στο εσωτερικό της ζώνης. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις προς το Συμβούλιο και δεν έχει νόημα να ζητάμε τώρα από τα κράτη-μέλη να κάνουν μέσα σε ένα χρόνο 20 μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι ανέφικτο και ανόητο. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι θα πρέπει τρεις μεγάλες ανά έτος, αλλά θα πρέπει όμως να υπάρχει μια εθνική προσπάθεια για την επίτευξη των μεταρρυθμίσεων αυτών, οι οποίες έχουν αρχικά προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Να πω τώρα δύο λόγια για το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί κατά τη διάρκεια της ε, προεκλογικής εκστρατείας εγώ ζήτησα μια δίκαιη συμφωνία για τη Βρετανία και είμαι πεπισμένος ότι θα έχουμε μια τέτοια συμφωνία. Εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, συνέστησα μια ειδική ομάδα για τις ε, διαπραγματεύσεις με τη Βρετανία υπό την ηγεσία μάλιστα ενός Βρετανού. Βρετανού πολίτη, ο οποίος είναι Ευρωπαίος. Ε, μα δεν είναι αντίφαση αυτό. Ε, ήμουν μεταξύ του Τζόναθαλ Φόλ και του Νάιτζελ Φάρατζ, τελικά διάλεξα τον ε, κύριο Φόλ και ο Νάιτζελ βεβαίω θα είναι ο μεγαλύτερο ε, υποστηρικτή του, γιατί ο ένα είναι Βρετανό και ο άλλο είναι Βρετανό και Ευρωπαίο. Οπότε νομίζω θα τα βρείτε. Λοιπόν, οπωσδήποτε το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βρετανική κυβέρνηση και η Βρετανή πολιτική έχουν δίκιο όταν ασκούν κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λένε ότι είναι γραφειοκρατική για την υπερβολική δόση ρυθμίσεων και κανονισμών σκοπεύει η Επιτροπή μου να μειώσει τους κανονισμούς. Και μάλιστα ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο Φρανς Τίμερμανς και εγώ καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να έχουμε καλύτερη ποιότητα κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως δεν σημαίνει καταστροφή, ούτε σημαίνει έλλειψη κανόνων. Ούτε σημαίνει πως ε, θα πρέπει να απέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα πράγματα τα οποία πρέπει να οργανωθούν στην Ευρώπη. Ξεκινήσαμε την ε, ψηφιακή ενιαία αγορά, την ενεργειακή ένωση. Βήμα-βήμα, σιγά-σιγά ολοκληρώνουμε την εσωτερική αγορά. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι αιτήματα της ε, Βρετανικής κυβέρνησης και κυρίως ε, και των ε, Βρετανών πολιτικών και όσων χαράζουν πολιτική. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά δεν μπορεί να τα ζητάτε από αυτήν την Επιτροπή. Αυτή η Επιτροπή αυτά ακριβώς κάνει. Και θα ήθελα οι Βρετανοί φίλοι μας να στηρίξουν την ε, πρωτοβουλία της Κομισιόν σε αυτόν τον τομέα. Το ίδιο ισχύει δε και για την ανάγκη που διαπιστώνουμε ε, για να συναυθούν εμπορικές συμφωνίες με πάρα πολλά κράτη του κόσμου μεταξύ των οποίων και η Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων. Εγώ είμαι υπέρ της συμφωνίας TTIP όπως λέγεται. Αλλά δεν είμαι υπέρ του να μην έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες, ευρωπαϊκές αρχές. όπως και στην περίπτωση της Βρετανίας. Η ελεύθερη ε, διακίνηση των εργαζομένων δεν μπορεί να παραβιαστεί. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για την διατλαντική αυτή συμφωνία. Έχουμε κάποιες βασικές αξίες και αρχές οι οποίες δεν είναι δυνατόν να παραβιαστούν κατά τη διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ. Και, όπως ε, και η Σεσίλια Μάνστρομ, η Επίτροπος Εμπορίου που έχουμε, είμαι υπέρ της μέγιστης διαφάνειας. Αλλά δεν είναι δυνατόν οι διαπραγματευτικές θέσεις να χαράζονται δημοσίως. Δεν είναι δυνατόν να λέμε το τι σκοπεύουμε να κάνουμε και ποιες είναι οι θέσεις αναδίπλωσης και τι θα κάνουμε σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτές οι απόψεις μας. υπάρχει η διαφάνεια, αλλά υπάρχει και η σοβαρότητα. Και οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνονται με τρόπο σοβαρό. Να πω και κάτι για την Ουκρανία. Εμείς στηρίζουμε τις ε, προσπάθειες του Προέδρου της ε, Ουκρανίας και πρέπει να τον ε, στηρίζουμε γιατί έχει το θάρρος ε, της γνώμης του και βεβαίως κάνει τα όσα πρέπει να γίνουν. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Και όσοι αμφιβάλλουν για την ε, εμπλοκή μας στην ε, Ουκρανία θα αποδειχθεί ότι κάνουν λάθος. Γιατί σε όλες τις συνομιλίες με τον πρόεδρο Ποροσέγκο ανταποκριθήκαμε σε όλα τα αιτήματα της ε, Ουκρανίας και μάλιστα δώσαμε και 3,51 δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομική βοήθεια. Ήμασταν έτοιμοι για μια σαλίση της προμήθειας φυσικού αερίου της Ουκρανίας για το χειμώνα και συμβουλεύουμε και τους φίλους μας εκεί πέρα για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Θα καταβάλω λοιπόν κάθε προσπάθεια για να δώσω την δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει την δυνατότητα στους Ουκρανούς πολίτες να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση διαβατηρίων. Εάν ε, πληρούνται οι όροι, αυτό πρέπει να γίνει. Όπως είπε και ο Γκίφερ Χόφστατ πριν από λίγους μήνες σε αυτή την αίθουσα, οι αξίες του Μαϊντάν δεν αφορούσαν μόνο την ε, δημοκρατία και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι άνθρωποι εκεί που ζουν στην Ουκρανία δεν θέλουν μια χώρα διεφθαρμένη όπως είναι σήμερα η Ουκρανία. Οι Ουκρανοί δημοκράτες θέλουν μια χώρα χωρίς διαφθορά. Και σκοπεύουμε να τους βοηθήσουμε. Θα ήθελα να πω, επειδή τα παρακολουθώ αυτά τα ζητήματα, συνεχώς. Οι χώρες ε, μέλη οι ανατολικές, ειδικά των ε, Βαλκανίων, πρέπει να γνωρίζουν πως η ασφάλεια και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραβίαστα και πρέπει να το γνωρίζουν αυτό στη Μόσχα. Να το γνωρίζουν τα κράτη-μέλη και ειδικά των Βαλκανίων πως η ελληνική δεν είναι μια κενή λέξη. Είμαστε εκεί και θα είμαστε εκεί εάν χρειαστεί τα Βαλκάνια, η Πολωνία και άλλες χώρες. Κυρίως η Πολωνία και τα Βαλκάνια βεβαίως. Ναι. Όχι, όχι, δεν μπέρδεψα τις βαλτικές χώρες με τα Βαλκάνια, μην ανησυχείτε. Είναι, είναι πάρα πολύ ε, σημαντικές χώρες και να ξέρετε πως θα είμαστε εκεί εάν απειληθούν τα σύνορά τους. έχουμε υποχρέωση να τις προστατεύσουμε εάν χρειαστεί. Τι, για το στρατό του Λουξεμβούργου μιλούσατε. Ε, είναι εξαιρετικό στρατός. «771 στρατιώτες του Υπουργού συμπεριλαμβανομένου. Ε, δεν θα βοηθήσει πολύ ο στρατό του Λουξεμβούργου, αλλά θα βοηθήσουν οι άλλοι αν χρειαστεί. Ναι, ναι, καλά, καλά. Μα αναρωτιέμαι γιατί μου αρέσουν τόσο πολύ οι διακοπές σας. Τέλος μου αρέσει να με διακόπτετε, γιατί με εμπνέετε. Γιατί ε, μου θυμίζουν τι θα έπρεπε να σας έχω πει. Δεν θα ξεχάσω την συνάντηση που είχαμε τον ε, Νάιτζελ Φάρατς και την ε, ομάδα του. Ήταν πραγματικά πολύ ανοιχτή και ειλικρινής. Και πραγματικά βεβαίως αυτό είναι το μόνο κοινό μας ε, σημείο, το χιούμορ. Ε, κάτι είναι και αυτό, ναι. Έχω την άδεια του Προέδρου να μοιράσω το κείμενο για την κλιματική αλλαγή, γιατί είναι σημαντικό. Γιατί μιλάω ήδη 72 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα βλέπω. Και δεν θέλω κι άλλο, κι άλλο. Εντάξει. Έχω νέους φίλους λοιπόν. Αυτοί εδώ πέρα στο κέντρο ε, έχουν αρχίσει να κουράζονται. Εκεί στα ορεινά όμως θέλω να συνεχίσω. Ο πρόεδρος. Περιμένετε παρακαλώ μια στιγμή κύριε πρόεδρε της Επιτροπής. Ο βουλευτής στην θέση 358 έβαλε μια μάσκα με την ε, κυρία Μέρκελ. Κοιτάξτε, δεν την ε, αγαπάω ιδιαίτερα, αλλά βλέπω πως ε, έχει ομορφήνει. Νομίζω πως είναι ο κύριος Μπονάνο. Εντάξει κύριε Μπονάνο, κάνατε την παράστασή σας, καθίστε τώρα κάτω πάλι. Συνεχίστε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Μάλιστα. Όλα αυτά τα πληρώνει ο Ευρωπαίος Φορολογούμενος. Παρακαλώ κύριε Γιούγκερ. Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είναι ένα μέρος στο οποίο μπορεί να συναντήσει κανείς τα πάντα, τι να πω. Union in Ενωμένη στην διαφορά. Θα ήθελα τώρα να πω λίγα λόγια, μια και ο χρόνος πιέζει, για την κλιματική αλλαγή. Θα μοιραστεί το κείμενο της ομιλίας μου τις επόμενες ώρες. Απλά θα ήθελα να πω πως θεωρώ πως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ φιλόδοξοι ως Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς ε, οδεύουμε προς την διάσκεψη των ε, Παρισίων. Κάνουμε, νομίζω, σοβαρές προσπάθειες. Αντιμετωπίζουμε τις αιτίες της, ε, του επόμενου μεταναστευτικού κύματος, τις επόμενες δεκαετίες με το να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής. Γιατί αύριο θα έχουμε κλιματικούς πρόσφυγες και δεν θα πρέπει να εκπλαγούμε όταν τους δούμε. Πρέπει να δράσουμε τώρα. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Γι' αυτό θέλω η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξοι καθώς πλησιάζουμε προς ε, την διάσκεψη των Παρισίων. Θα ήθελα όμως να πω πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υπογράψει όποια συμφωνία να είναι. Η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι μια φιλόδοξη, εύρωστη και δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία. Αυτό είναι το καθήκον μας. Πρέπει να παλέψουμε γι' αυτό και να υψώσουμε τη φωνή μας κατά όσων διαφωνούν με κάτι τέτοιο. Η Ευρώπη δεν είναι ουδέτερη όταν μιλάμε για την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να είναι ένα παράδειγμα, υπόδειγμα για όλους τους άλλους. Ιδού κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. όχι η συνολική κατάσταση της Ένωσης αλλά δεν θέλησα να κάνω ποιητική περιγραφή της Ένωσης αλλά να περιγράψω με ένα λόγο που δεν θα τον πω στο σύνολό του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε καλή κατάσταση και νομίζω επίσης ότι καθήκον μου είναι κάτι να κάνω μπροστά σε όλους εκείνους που κατηγορούν την Ένωση. Προτείναμε ήδη ορισμένες ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις εγκρίναμε ένα πρόγραμμα για την μετανάστευση και δεν δέχομαι να, λέτε, να λένε ότι η Κομισιόν δεν έκανε τίποτα για τη μετανάστευση. Επίσης στη γερμανική τηλεόραση άκουσα υπουργού βαβαρούς να επικρίνουν την Κομισιόν για απουσία. Ήμουν διακοπές, ναι ήμουν, εσείς δεν πήγατε. Εγώ δέκα μέρες διακοπές που πήγα, τέσσερις από αυτές δούλεψα για την Ελλάδα και τις υπόλοιπες για την μετανάστευση. Από το Μάιο ήδη κάναμε προτάσεις. Τι να ανακαλύπτουμε τώρα το πρόβλημα της μετανάστευσης. Ανακαλύπτουν τώρα μόνο. Εμείς το ξέραμε. εγκρίναμε και άλλα συνοδευτικά μέτρα για την εσωτερική αγορά, για την ενέργεια για την κεφαλαία αγορά και μαζί με τους επιτρόπους για τη συνεργασία με τους οποίους χαίρομαι ιδιαίτερα. Όσοι από εσά υπήρξατε πρωθυπουργοί ξέρουν ότι η συνεργασία σε μια εκτελεστική και μια κυβέρνηση δεν επιτυγχάνεται εύκολα εγώ είμαι περήφανος για την Επιτροπή της οποίας προεδρεύω, διότι από τους πρώτους μήνες της εντολής μας, της θητείας μας, μπορέσαμε να υποβάλουμε στους δύο νομοθέτες μεγάλα σημαντικά νομοθετήματα και μεταρρυθμίσεις και τις δέκα προτεραιότητες για τις οποίες είμαι ιδιαίτερα περήφανος. Δεν είναι βέβαια ίσως όλα τέλεια, δεν ζούμε στον καλύτερο δυνατό κόσμο και επειδή δεν είναι κανείς τέλειος θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Εγώ ξέρω τις αδυναμίες της Ευρώπης αλλά ξέρω και τις τεράστιες αδυναμίες που θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε η Ένωση. Επομένως, μην θα συνεχίσουμε την προσπάθεια όσοι είστε πεπισμένοι Ευρωπαίοι. Σας ευχαριστώ κύριε Γιούνκερ Κυρίες και κύριοι, κύριε Γιούνκερ να σας πω κάτι. Γνωρίζουμε όλοι πως την προηγούμενη Κυριακή απεβίωσε η μητέρα σας. Και ο πατέρας σας νοσηλεύεται. Το ότι σήμερα λοιπόν βάλατε το καθήκον σας ε, πάνω από τα προσωπικά σας ε, συναισθήματα είναι κάτι το αξιοθαύμαστο και θα ήθελα να σας ε, ευχηθώ να σας διαβιβάσω τα συλληπιτήρια του σώματος για τον θάνατο της μητέρας σας. E τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Βέμπερ για το ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ακούσαμε από τον Πρόεδρο της Κομισιόν μια ανάλυση για την κατάσταση και σαφείς ε, προτάσεις. Και σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε από το πιο επίγον θέμα, την μεταναστευσή στο Μιλάνο που πήγαμε, συναντήσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Άλφανο και μας είπε μία ιστορία. Επισκέφθηκε ένα κέντρο φιλοξενίας ε, προσφύγων στο νότο της Ιταλίας, μίλησε με τη μητέρα, ε, η οποία μας είπε ότι ξεκίνησε από την Αφρική με πέντε παιδιά και έφτασε στην Ιταλία με ένα ζωντανό μας είπε πως η γυναίκα κοιτούσε το κενό. Γι' αυτό όταν μιλάμε για αριθμούς να σκεφτόμαστε πως ε, πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι και ο καθένας θα πρέπει να ανταποκριθεί στα ανθρωπιστικά του αισθήματα. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που χτυπάνε την πόρτα μας να εγγυηθούμε αυτή την βοήθεια και όπως ε, λέει ο κύριος Πρόεδρος όταν το καταφέρουν φτωχές χώρες όπως ο Λίβανος και η Ορδανία θα πρέπει να το κάνει και η Ευρώπη. Ακούσαμε λοιπόν διάφορες δηλώσεις. Θα ήθελα να σας πω, π.χ. ο κύριος ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός θέλει να πάρει μόνο μη μουσουλμάνους, μόνο χριστιανούς. Και Πρέπει να το πούμε αυτό, εμείς οι χριστιανοδημοκράτες δεν είμαστε υπερήφανοι στην Ευρώπη ε, το ότι, για το ότι εφήβραμε δικαιώματα για τους χριστιανούς. Είμαστε περήφανοι για το ότι εφήβραμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, βλέπουμε πως η Ευρώπη απέτυχε. Το διαβάζουμε παντού έδωσα μια συνέντευξη στην Κοριέρα ε, Ντελασέρα και εκεί πέρα ακριβώς ο Φράνκο Φρατίνη μου υπενθύμησε πως πριν από 10 χρόνια είχε στείλει ένα email με την έννοια του τρίτου ασφαλούς κράτους και δεν πέρασε αυτή η πρόταση. Αυτό το οποίο λοιπόν αποτυγχάνει δεν είναι η Ευρώπη. Βλέπουμε τις προτάσεις της Κομισιόν, δεν αποτυγχάνουν οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Αποτυγχάνει ο εθνικός εγωισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρόλα αυτά πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα. Δύο τρίτα των ανθρώπων που μπήκαν στην Ευρώπη πέρσι απελάθηκαν. Οπότε τίθεται το ζήτημα της απέλασης, της ε, προστασίας αλλά και των ασφαλών τρίτων χωρών. Πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε την κατάχρηση του συστήματος. Κυρίες και κύριοι, έχουμε λοιπόν την ε, μετανάστευση. Υπάρχει και το άλλο τεράστιο θέμα, η οικονομική κατάσταση της υπήρου μας. Χρειαζόμαστε θέσεις εργασίας, χρειαζόμαστε ένα οικονομικό μέλλον για τους νέους μας. Αναφέρθηκε η εσωτερική αγορά. Μέχρι στιγμής πάντα δημιουργούσε ανάπτυξη και ευημερία. Χρειαζόμαστε ελεύθερο εμπόριο. Δεν μας αφαιρεί κάτι το ελεύθερο εμπόριο. Αντιθέτως πάντα μας βοηθούσε. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την ανεργία των νέων. Υπάρχει και το πακέτο της κινητικότητας της ε, Κομισιόν και όσον αφορά τους αγρότες θα ήθελα να πω πως τους στηρίζουμε και οπωσδήποτε θα δώσουμε τη σωστή κατεύθυνση στην κοινή οργάνωση αγοράς. Τέλος, αν μου επιτρέπετε κάτι για την κατάσταση στην Ελλάδα. Όποιος θέλει να δει πώς πάνε τα πράγματα σωστά πρέπει να δει την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και τις άλλες χώρες. Όποιος κοιτάει όμως την Ελλάδα βλέπει πως ε, πέρασαν οι χαμένοι μήνες και είχαμε εδώ πέρα μια συζήτηση με τον κύριο Πρωθυπουργό σε αυτή την ε, αίθουσα, τον κύριο Τσίπρα, αλλά πρέπει να πω πως ε, αξίζει σεβασμό η αλλαγή πορείας ε, που έκανε γιατί χωρίς μεταρρυθμίσεις δεν έχει μέλλον η χώρα του και έτσι απέδειξε ο κύριος Τσίπρας πως η αριστερή ιδεολογία απέτυχε σε αυτή την Ήπειρο γι' αυτό και υποχωρούν και υποδέμω στην Ισπανία. Υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να πούμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το ζήτημα της ε, Ουκρανίας. Ε, αναφέρθηκε το ζήτημα της βίζας ε, θα πρέπει να δούμε το τι θα γίνει με ε, την κατάπαυση του πυρός. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούμε την κατάσταση που θέλει ο Πούτιν, μια παγωμένη σύγκρουση. Τέλος, ε, για τις προτάσεις Μεγάλης Βρετανίας, οπωσδήποτε είμαστε άνοιχτοι και θα συμμετάσχουμε στην συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα χρόνο επιτροπή του Ζαν Κλουτ Πρόκειται για μια πολιτική επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, επικεντρωθήκατε στα ουσιαστικά ζητήματα καταφέρατε να έχουμε μια πολιτική προσέγγιση και βεβαίως ε, το ωραιότερο νούμερο είναι το 1,65 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν σε αυτήν την Ήπειρο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Εξαγγείλατε ένα προεκλογικό πρόγραμμα, το υλοποιείτε και η ομάδα μας θα σας στηρίξει. Για τους Σοσιαλδημοκράτες έχει ο κύριος Πιτέλα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βλέπω ότι η θέση του Προέδρου του Συμβουλίου είναι κενή. Ρητορικά το λέω βέβαια αλλά αναρωτιέμαι ε, ποια είναι η αιτία για τις καθυστερήσεις ε, οι οποίες δημιουργούνται όταν πρέπει να δώσει η Ευρώπη κάποιες απαντήσεις. Εσείς κύριε Γιούνκερ είστε παρόν ε, και όπως το θύμισε ο πρόεδρος Σούλτς ήρθε εδώ και είστε βαθιά λυπημένος αλλά παρόλα αυτά με την παρουσία σας και με την ομιλία σας δείξατε ότι αγαπάτε τα ευρωπαϊκά όργανα. Σας ευχαριστώ γι' αυτό, σας ευχαριστώ και για την εξαιρετική ομιλία σας. Και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι ειλικρινής όπως εσείς και για τα θέματα της μετανάστευσης όπως είπατε η Ευρώπη πρέπει ένα πράγμα να κάνει, να είναι η Ευρώπη. Να θυμηθεί η Ευρώπη ότι βασίζει την δημιουργία της στις αρχές της αλληλεγγύης και στους πρόσφυγες μετά τον πόλεμο η Ευρώπη δεν υπάρχει σαν κοινότητα χωρίς αλληλεγγύη. Θα δείτε ποια είναι η αλληλεγγύη που επιδεικνύουν οι Ευρωπαίοι πολίτες καθημερινά. Κατεβείτε στους δρόμους και θα δείτε πώς βοηθούν οι απλοί πολίτες. Λοιπόν, η Ευρώπη θα πρέπει στην ουσία να μάθει από το λαό της. Δεν θα πρέπει να είμαστε δειλοί πάνω σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει θετικά πράγματα στον τομέα της μετανάστευσης. Οι προτάσεις της για την κατανομή των προσφύγων είναι σωστές προτάσεις. Οι προτάσεις της για το Δουβλίνο είναι σωστές προτάσεις. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο το κατεπήγον εδώ. Υπάρχει ένα κοινωνικό πρόβλημα. Σε αυτή την Ήπειρο στην ουσία σιγά σιγά έχει ξεκινήσει μία σιωπηλή αποσχιστική τάση που διαιρεί τους πλούσιους από τους φτωχούς. Μιλήσατε για το κοινωνικό 3α. Παρακαλώ θα ήθελα οι κανόνες που ισχύουν να εφαρμόζονται, να εφαρμόζονται σωστά και να καταδικάζονται οι καταχρήσεις. Θα πρέπει να καταδικαστεί το κοινωνικό dumping. Απαιτείται μια αλλαγή στην οδηγία για την ε, απόσπαση των εργαζομένων και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις φοβερές αυτές συμβάσεις μηδενικού ωραρίου. Θα πρέπει να πληρώνονται οι φόροι εκεί όπου παράγεται το κέρδος. Αυτό σημαίνει δηλαδή μια κοινή φορολογική βάση και ένα reporting αναχώρα, έκθεση αναχώρα. Και να μην ξεχνάμε αυτό που συνέβη στην Ελλάδα, δεν το ξεχάσατε κι εσείς. Η οικονομική αυτή ένωση και κοινωνική ένωση δεν λειτουργεί σωστά πρέπει ακριβώς να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατόν η έκθεση των πέντε προέδρων όταν δημοσιευθεί. Θα πρέπει επίσης να μην ξεχνάμε και τις προτάσεις της Περβάνς Μπερές που ενέκρινε η Ολομέλεια. Να υπάρξει φορολογική επίσης ε, ε, δικαιοσύνη στον τομέα της φορολογίας. Υπάρχει η μάστιγα ε, του δημοσίου χρέους. Λοιπόν, το ξεχνάμε αυτό, όχι. Ας μιλήσουμε για ευρωομόλογα. Ας μιλήσουμε για επενδύσεις που θα στηρίξουν με πραγματικούς τρόπους την ευρωπαϊκή κοινωνία. Μια κοινωνία με μια οικονομία η οποία είναι κυκλική και θα πρέπει να γίνει βιώσιμη. Και εδώ δεν ξεχνάμε και για το περιβάλλον της συνάντηση στο Παρίσι. Ε, ο πόλεμος κύριε Σούλτς είναι στις πύλες της Ευρώπης, Συρία, Λιβύη, ε, εν μέρη και στην Ουκρανία. Αλλάζει η εξωτερική πολιτική. Ευχαριστούμε την ε, Φεντερίκα Μογκερίνη στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Έχουμε κάνει βήματα πρόοδου, έχουμε μια παρουσία αναγνωρισμένη που εκτιμάται σωστά βέβαια, τα προβλήματα υπάρχουν υπάρχουν γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε βάθος τις αιτίε που γεννούν τις σειράξεις αυτές. Πρέπει λοιπόν να επιστρέψουμε στις βασικές μας αξίες, πρέπει να επενδύσουμε στην Αφρική πολιτικά και σε επίπεδο βοήθειας με μακροπρόθεσμη προοπτική. Δεύτερη ευκαιρία, συμφωνείτε κύριε Γιούνκερ με μένα, δεν θα έχουμε η Ευρώπη πρέπει να επιστρέψει στην δημοκρατία και να καταδικάσει τον ηγεμονισμό της αγοράς και την αγοραία αντίληψη για την οικονομία. Δεν πρέπει να είμαστε διστακτικοί σε αυτό. Θα πρέπει να μας θυμούνται οι επόμενες γενιές όχι σαν αυτοί που διαχειρίστηκαν την ύφεση και την πτώση αλλά σαν αυτούς που άλλαξαν την πορεία της Ευρώπης. E Ευχαριστώ για το ECR ο πρόεδρος ο κύριος Καμάλ. Κύριε Γιούνκερ, καταρχάς θα ήθελα να επαναλάβω και εγώ αυτά που είπε ο Μάρτιν Σούλτς, δηλαδή να σας αποτίσω ένα φόρο τιμής για το θάρρος σας που προσήλθατε σήμερα λόγω της υψηλής σας αίσθησης καθήκοντος. Δεν, δεν σας προετοιμάζω επίθεση, μην ανησυχείτε. Χρόνο με το χρόνο ακούμε πολλά παχιά λόγια εδώ μέσα. Ακούμε πολλά ιδεολογικά πράγματα, ιδεαλισμό. Μας λένε μόνο η Ευρώπη είναι απάντηση. Άλλοι λένε ότι η Ένωση είναι η πηγή του προβλήματός μας. Γι' αυτό δεν γίνεται τίποτα ποτέ. Γι' αυτό η Ένωση αντιμετωπίζει συνεχείς κρίσεις. Ξέρω ότι πολλοί από εμά από όλε τι πολιτικές ιδεολογίε γίναμε πολιτικοί γιατί θελήσαμε να βοηθήσουμε. Εδώ παραλύουν όλες οι συζητήσει με δογματικό και ιδεολογικό τρόπο. Είναι κάστρα στην άμμο όλα αυτά. Άλλες φορές η συζήτηση γίνεται φαρσοκομωδία όπως όταν ο συνάδελφος ήρθε με μάσκα της Μέρκελ, κατέβηκε. Η κρίση των προσφύγων όμως είναι ένα από τα σοβαρότερα παραδείγματα που χρειάζονται αντιμετώπιση. Πολλοί εσκεμένα θέλουν να υπάρξει σύγχυση μεταξύ προσφύγων και μεταναστών. Είτε να τους φέρουν όλους μέσα είτε να τους κρατήσουν όλους απ' έξω. Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι πρόκειται για ανθρώπους που ζητούν άσυλο, είναι αυτοί είναι πρόσφυγες. Ξέρουμε από τι θέλουν να διαφύγουν. Αλλά υπάρχουν και άλλοι. Είναι φυσικό να θέλουν όλοι να βρουν μια καλύτερη ζωή. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι θα ακολουθηθούν οι σωστοί κανόνες. Υπάρχει παράνομη μετανάστευση σήμερα και πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτή. Επίσης όμως πρέπει να εξηγήσουμε στους εκλογείς μας ότι οι σειράξει στην Ερυθρέα, την Ουκρανία, τη Λιβύη, τη Συρία θα κρατήσουν πολύ καιρό. Αυτοί που λένε ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις απλώς ψεύδονται. Στην Ένωση όμως αντί να ψάξουμε κοινέ λύσεις βλέπουμε χώρες και θεσμούς που απλώς προσπαθούν να βρουν ένα αποδιοπομπαίο τράγο αντί να ψάχνουν λύσεις. Μερικές χώρες ξαναγράφουν τους κανόνες μόνες τους. Άλλες τους παραβιάζουν. Αλλά η Ένωση θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμη για τη συνεργασία των χωρών μεταξύ τους ώστε να βρεθούν κοινέ λύσεις. Ας καθίσουμε λοιπόν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων και δεν εννοώ μόνο τις δικές μας χώρες. Είναι διεθνής η κρίση. Χρειάζεται διεθνής ανταπόκριση. Από τους πρόσφυγες της Συρίας το 90% έχουν καταρχήν πάει στο Λίβανο, την Ιορδανία και την Τουρκία. Άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής όμως αρνούνται τους πάντες. Να είναι σαφές. Το να λέμε στις χώρες τι πρέπει να κάνουν, το να επιβάλλουμε σχέδια δεν οδηγεί πουθενά. Μπορεί να ευκολύνει ορισμένους για τις συνειδήσεις τους, αλλά δεν είναι λύση, διότι Διαφορετικές χώρες μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς με διαφορετικό τρόπο. Μερικές μπορεί να θέλουν όντως μετανάστες, επιλογή τους είναι. Άλλες θα πούν ότι θέλουν να βοηθήσουν ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους. Έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε τα εκατομμύρια αυτών των ανθρώπων. Όχι μόνο μερικές χιλιάδες που καταφέρνουν να φτάσουν μέχρι τις χώρες μας. Και γι' αυτό μερικές χώρες όπως και η δική μου επικεντρώνουν την προσοχή τους στο θέμα των καταβλισμών προσφύγων και δίνουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ στην ε, διοργάνωση, καλύτερη διοργάνωση των καταβλισμών αυτών ήδη στη Μέση Ανατολή και προσπαθούν να βελτιώσουν τις υποδομές επιτόπου. Άλλες χώρες επίσης μπορούν να συμβάλλουν με περισσότερα χρήματα και βοήθεια να οργανώσουν κέντρα υποδοχής ή αδειοδότησης κοντύτερα στις πηγές της μετανάστευσης. Άλλες μπορούν να καταπολεμήσουν τους δουλεμπόρους, αλλά όλοι μαζί με μεγαλύτερη επένδυση σε πόρους μπορούμε να διαχωρίσουμε και όσους είναι πράγματι πρόσφυγες από εκείνους που δεν είναι. Πρέπει να υπάρχει ρεαλιστική ανταπόκριση χωρίς ιδεολογίες. Πρόεδρε Γιούνκερ, εδώ και ένα χρόνο είδαμε φοβερή πίεση επί της Ευρώπης, όχι μόνο την κρίση της Ευρωζώνης αλλά και τους πρόσφυγες. Πρέπει να βρούμε λύσεις ρεαλιστικές. Τελείωσε πια η εποχή που θα κουνάμε μόνο το δάχτυλό μας βρίσκοντας ενόχους. Να καθίσουμε λοιπόν όλοι μαζί κάτω στο τραπέζι και να βρούμε μια λύση. Δεν χρειαζόμαστε νέο σιδηρούν παραπέτασμα αλλά σιδηρά θέληση για αντιμετώπιση της κρίσης. Ελπίζω να με ακούσετε. Ευχαριστώ για τους φιλελεύθερους τώρα ο κύριος Φερχόφστατ. Πρώτα απ' όλα κύριε Πρόεδρε, σας συλληπήθηκα και προσωπικά βεβαίως. Θα ήθελα τώρα να σας ε, διαβιβάσω και τα συλληπιτήρια ολόκληρης της ε, ομάδας μου. Κύριε Πρόεδρε, ίσως του χρόνου να ε, γίνει διαφορετικά η συζήτηση και να προσκαλέσουμε και τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων εδώ πέρα ε, νομίζω υπάρχει χώρος στα έδρανα γιατί δεν ξέρω ο κύριος Γιούνκερ αν έχει 90 λεπτά να μιλήσει στο Συμβούλιο και μετά να δώσουμε και την δυνατότητα στον ε, κύριο Τούσκ να είναι εδώ πέρα γιατί δεχτήκαμε να υπάρχει μόνιμος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε πρέπει να είναι εδώ και ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Είναι στη Μέση Ανατολή, στη Ραμάλα, την Ιερουσαλήμ ε, και πηγαίνει ε, όμως να έπρεπε να είναι σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου. Αλλά ας έρθουμε λίγο στην ουσία του προβλήματος. Η ουσία είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης και ενότητας μεταξύ των κρατών μελών, κύριε Καμάλα. Αυτό το οποίο υπερασπίζεται εδώ πέρα είναι το να διαλέγει κανείς τους πρόσφυγές του. Ναι, η Βρετανία το κάνει έτσι, η Γερμανία αλλιώς, η Ουγγαρία οπωσδήποτε αλλιώς, όπως ξέρουμε. Μα δεν αντιμετωπίζονται έτσι αυτά τα ζητήματα. Η κρίση αυτή είναι συλλογική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό διακυβεύεται και πρέπει να σταματήσουμε να αντιδρούμε. Τι έγινε λοιπόν, τον Απρίλιο εμφανίστηκε η κρίση, αυξήσαμε λίγο τον προπολογισμό της Frontex και νομίζαμε ότι λύθηκε. Δεν λύθηκε. 50 μήνες μετά έφτασαν όλοι αυτοί στο τούνελ της ε, Βρετανίας και τι κάνουμε, ε, λίγα λίγα περισσότερα χρήματα για σκηνές και λεφτά. Και άρα λύθηκε το πρόβλημα στο καλέ, τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Μετά, η Βουδαπέστη, αυτά τα οποία βλέπουμε, απίστευτα. Στο σταθμό του τρένου να συσσωρεύονται, τους μεταχειρίζονται χωρίς κανένα σεβασμό και μετά λέμε ας ανοίξουμε λίγο τα τρένα να πάνε στην Αυστρία και άρα το ξεφορτωθήκαμε το πρόβλημα. Όχι, είναι πραγματικά ντροπή αυτή η αντιμετώπιση. Δεν μεταχειριζόμαστε σωστά τους πρόσφυγες. Πρέπει να αναγνωρίσουμε κάποιες ε, χώρες ε, ανέλαβαν την ευθύνη τους. Η Γερμανία, παραδείγματος χάρη, στο Μόναχο δέχτηκαν 20.000 ε, άτομα σε 5 μέρες. Ε, άλλες λένε εμείς θα πάρουμε τόσο σε 5 χρόνια και άλλες λένε όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Και ευτυχώς πρέπει να πούμε υπάρχουν χιλιάδες απλοί άνθρωποι που επέδειξαν αλληλεγγύη, περισσότερη αλληλεγγύη από τους ε, ηγέτες μας. Οπότε το μήνυμά μου. Όχι προς εσάς κύριε Γιούνκερ, αλλά ειδικά προς ε, το Συμβούλιο είναι να σταματήσουμε να λέμε ότι είναι κρίση της Ευρώπης. Δεν είναι κρίση της Ευρώπης. Είναι κρίση έλλειψης Ευρώπης. Ας το πούμε αυτό το πράγμα. Το Δουβλίνο δεν είναι η Ευρώπη, είναι η άρνηση της Ευρώπης. Να λέμε, α, ας την πληρώσουν οι Έλληνες και οι Ιταλοί. Γι' αυτό ακριβώς το Μάιο ήδη κάνατε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για να μοιραστούμε το βάρος και ελπίζω το Συμβούλιο σε λίγες μέρες και όχι μήνες να δεχτεί κάποιες από αυτές τις ε, προτάσεις και ίσως να υπάρχει και ένα νόμιμο σύστημα μετανάστευσης γιατί λένε πως δεν είναι το ίδιο οι, μετανα... δεν είναι το ίδιο οι πρόσφυγες και οι οικονομικοί μετανάστες. Ναι το ξέρουμε αλλά πρέπει να υπάρχει ένα νόμιμο σύστημα μετανάστευσης. Ένα, όχι 28 όπως υπάρχουν σήμερα, όπως έχουν οι Αμερικάνοι την πράσινη κάρτα. Έχουμε και εμείς μπλε κάρτα αλλά η μπλε κάρτα είναι το 21 ο σύστημα μετά τα 28 και μόνο η Γερμανία το χρησιμοποιούσε. Πρέπει να αλλάξει λοιπόν αυτό και χαίρομαι για το ότι ανακοινώσατε ότι το 2016 θα προτείνεται ένα σύστημα νόμιμης μετανάστευσης. Και τέλος, το πιο σημαντικό νομίζω κύριε Πρόεδρε είναι πως δεν μπορούμε να αποφύγουμε μια τέτοια κρίση. Πάντα θα πληρώνουμε το τίμημα. Μην νομίζετε ότι μπορεί να υπάρχει σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, στο κέρας της Αφρικής και να λέμε όχι είναι μακριά από την Ευρώπη. Εμείς το πληρώνουμε και είμαστε πεπισμένοι πως ο πόλεμος στη Συρία δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Ε, ολοκάναμε συζητήσεις και λέγαμε «Α, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα για να βοηθήσουμε τις δημοκρατικές δυνάμεις». Δημιουργήσαμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ήρθε το Ισλαμικό κράτος και δεύτερον μια τεράστια προσφυγική κρίση. Οπότε νομίζω πως κάτι πρέπει να κάνουμε. Εάν το συμπέρασμα είναι να επαναλαμβάνει ο καθένας την αποψή του εδώ μέσα, δεν αρκεί. Χρειάζεται μια νέα πρωτοβουλία και θεωρώ πως στο πλαίσιο του ΟΗΕ ε, πρέπει να τελειώσει η αιματοχυσία στη Συρία, να σταματήσει η τρομοκρατία, να είναι ξανά ασφαλή χώρα η Συρία για να μπορέσουν να επιστρέψουν κάποτε οι πρόσφυγες. Οπότε η έκκλησή μου προς εσάς κυρία Μογκερίνη και προς ε, τον πρόεδρο του Συμβουλίου είναι εσείς να ζητήσετε από τους εκπροσώπους μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να ξεκινήσουν μια νέα πρωτοβουλία το συντομότερο δυνατόν. Αυτή είναι η μόνη λύση. Σας ευχαριστώ. Για την Γκουε τώρα η κυρία Τσίμερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γιούνκερ και εξ ονόματος της δικής μου ομάδας να σας εκφράσω τα συλληπιτήριά μας. Σας διαβεβαιώ πως ε, πραγματικά συμπάσχουμε με τον άνθρωπο Ζαν Κλοντ Τώρα για την ομιλία που εκφωνήσατε για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το πρόβλημα της ε, μετανάστευσης. Να πω δύο πράγματα. Είναι γνωστό πως ο Δίας απήγαγε την Ευρώπη την πριγκίπισσα αυτή, η οποία ήταν νομίζω η πρώτη μετανάστης στην Ευρώπη. Μας έδωσε το όνομα αυτής της Υπήρου. Γι' αυτό λεγόμαστε Ευρωπαίοι. Εσείς είπατε πως ε, είναι ψευδέστηση να πιστεύουμε πως ε, το πρόβλημα αυτό θα λυθεί σύντομα. Πράγματι, είναι ψευδέστηση. Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του, ε, του αιώνα μας και θεωρώ πως ε, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε εξίσου σοβαρά όπως την κλιματική αλλαγή ως ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Τις ε, προτάσεις σας εγώ τις βλέπω ως μήνυμα, μήνυμα σε αυτούς είτε είναι εντός της αίθουσα είτε είναι υπεύθυνοι στα κράτη-μέλη, είτε λένε ανοιχτά ρατσιστικές θέσεις ε, και λένε πως η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι ανοιχτή, αλλά η Ευρώπη πρέπει πρώτα απ' όλα να φροντίσει τα δικά της συμφέροντα. Και επανέρχονται σε εθνικές και εθνικιστικές θέσεις. Να δούμε τις προτάσεις σας. Κάποιες μου φαίνονται ως ένα καλό βήμα. Κάποιε δεν πάνε αρκετά μακριά, αλλά νομίζω πως θα έχουμε την ευκαιρία να τις δούμε στην συζήτηση. Σε κάθε περιπτώση υποστηρίζω όλες τις προτάσεις που μιλάνε για νόμιμες δυνατότητες μετανάστευσης. Πως ε, πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη και αλληλέγγυα στάση και να μην παραμείνουμε σε μια ποσόστοση η οποία δεν θα λαμβάνει υπόψη τις ατομικές ανάγκες ε, των ανθρώπων, επανένωση οικογενειών κτλ. Πρέπει να ε, ληφθούν υπόψη αυτά. Και βεβαίως ε, σημειώνουμε αυτό το οποίο λέτε για την Σύμβαση της Γενέβης, για το δικαίωμα στο, στο άσυλο, ότι δεν θα μειωθούν αυτά τα δικαιώματα. Αυτά πρέπει να παραμείνουν. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι κατεπήγον για την Ελλάδα και για το πώς λύνουμε τα προβλήματα μας εντός Ένωσης. Ειδικά στο ζήτημα της Ελλάδας και των προσφύγων βλέπουμε ότι στέμνονται αυτά τα δύο πράγματα. Οι εικόνες από την ε, ΚΟ βλέπουμε πως ε, τίθενται ερωτήματα για το αν λειτουργεί καν ε, το κράτος και αν μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες του και απέναντι στους πρόσφυγες. Στην Ουγγαρία επίσης βλέπουμε πως ταπεινώνονται χώρες και επίσης είναι σαφές πως ε, οι Υπουργοί των ε, Οικονομικών πλέον ε, έχουν αναλάβει τη διακυβέρνηση της Ευρώπης. Οι αρχηγοί κρατών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν γίνει θεατές. Αυτά πρέπει να τελειώσουν και αν είμαστε σοβαροί θα πρέπει κάποια στιγμή οι αρχηγοί των κυβερνήσεων να φύγουν από την κοντόφθαλμη και εθνικιστική λογική τους γιατί θα καταστρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Τσίμερ, συντομεύετε. Ναι, ναι, μία λέξη ακόμα. Ο κύριος Γιούνκερ ε, μίλησε τρεις φορές παραπάνω ο κύριος Γιούνκερ. Λοιπόν, είπατε πως δεν πρέπει να μετράμε την κάθε λέξη. Δεν το έκανα στην ομιλία σας, αλλά κοίταξα ποιες είναι οι προτεραιότητές σας. Δεν μιλάτε για τα κοινωνικά, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο ως προτεραιότητα. Αλλάξτε το αυτό, αλλάξτε το. Αυτή είναι η κοινή μας αποστολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τσίμερ, το κάνετε συνεχώς. Είμαι πάντα γενναιόδωρος, μιλήσατε δύο λεπτά παραπάνω και μετά να μου λέτε πως ε, μίλησε παραπάνω ο κύριος Γιούνκερ, άρα μπορώ και εγώ. Ε, εντάξει. Δεν ε, είστε, σας παρακαλώ. Και από εκεί η μεριά δεν είστε εσείς στο χρονόμετρο του Κοινοβουλίου, δεν χρειάζομαι την βοήθειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Λάμπερτς. Ευχαριστώ. Κύριε Γιούνκερ, συμφωνώ μαζί σας. Στις δύσκολες στιγμές που ζείτε σήμερα βρίσκομαι κοντά σας, αλλά θα ήθελα να μπορώ να πω το ίδιο και για αυτά που κάνετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση βασίζεται στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελευθερίας, δημοκρατίας, κράτους δικαίου, καθώς και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και οι μειονότητες. Αυτές είναι οι κοινέ αξίες στα κράτη-μέλη σε κοινωνίες πλουραλισμού, ισότητας και όχι μυσαλλοδοξίας και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Αυτά πρέπει να συζητήσουμε σήμερα. Για ποια ένωση μιλάμε όταν η μόνη ανάπτυξη που υπάρχει στην Ευρώπη είναι η ανάπτυξη της ανισότητας και της ανέχειας και της ανεργίας ενώ τα κράτη-μέλη πολεμάνε το ένα το άλλο φορολογικά. Για ποια ένωση μιλάμε όταν μπροστά στο δράμα των προσφύγων μερικοί αρχηγοί κυβερνήσεων έχουν μόνο φραγμούς να προτείνουν. Για ποια ένωση μιλάμε όταν το Συμβούλιο γίνεται θέατρο των εθνικών ανταγωνισμών. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συνθήκη της Λισαβόνας μας μιλάει για συνεχώς στενότερη ένωση μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Παρ' όλα αυτά, η ένωση που αναφέρεται στο άρθρο 2 της συνθήκης είναι ζωντανή. Ζει μέσω όλων εκείνων που καταλαβαίνουν τη σημασία της ανθρωπιστικής και δημοκρατικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε και θέλουν να κάνουν κάτι από κοινού οι συμπολίτες μας που κάθε μέρα βρίσκουν καινούργιους τρόπους αντιμετώπισης της ανισότητας και σεβασμού της αξιοπρέπειας. Τους δασκάλους που δίνουν στα παιδιά μας τα εργαλεία για να δημιουργήσουν τη ζωή τους, τους γεωργούς που μας τρέφουν, τους ερευνητές που βρίσκουν σωστές και βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα της εποχής μας, στους επιχειρηματίες που βρίσκουν καινοτόμους τρόπους για να λειτουργήσουν, στους τραπεζίτες που θέλουν να εξυπηρετεί την κοινωνία η τράπεζα. Σε όλους όσους βρίσκουν τρόπους εναλλακτικής ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα. Επίσης σκέφτομαι εκείνους και εκείνες που αντιστέκονται στη δικρατεία του βραχυπρόθεσμου κέρδους και της εκμετάλλευσης του ανθρώπου και της φύσης. Σε αυτή την εποχή λοιπόν κύριε Πρόεδρε δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα ευρωπαϊκού πνεύματος από την υποδοχή προσφύγων από τους πολίτες σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίες και κύριοι είναι το αντίθετο του κλεισίματος στον εαυτό μας ότι έτσι αναπόφευκτα θα πολεμάνε ο ένας τον άλλον οι Ευρωπαίοι αν δεν γίνει σεβαστό αυτό το πνεύμα. Και με αυτούς τους συμπολίτες μας κύριε Γιούνκερ, κύριε και κύριοι πρέπει να οικοδομήσουμε συμμαχίες και να ξαναγεννηθεί η ελπίδα. Αλλιώς η Ευρώπη θα χαθεί μπροστά στην πρόκληση των μεταναστών και προσφύγων θυμηθείτε ότι ο Πάπας μας είχε πει εδώ μέσα ότι η Ευρώπη πρέπει να βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις με αλληλεγγύη. Και εσείς από νωρίς κύριε Γιούγκερ από την Άνοιξη λάβατε τέτοια μέτρα. Χρειάζεται μια νέα κλίδα κατανομής των προσφύγων. Μάλιστα γιατί είναι το, ο μόνος τρόπος να καταπολεμηθεί το business των δουλεμπόρων. Επίσης πρέπει να λάβουμε μέτρα άμεσης ανάγκης. Σας κάνω μια συγκεκριμένη πρόταση. Το κοινοβούλιο μας δουλεύει λιγότερο από 50 μέρες το χρόνο σε αυτή την αίθουσα. Υπάρχουν γραφεία με μπάνιο και με θέρμανση. Θα μπορούσαν αυτά τα κτίρια να διατεθούν προσωρινά για τους πρόσφυγες και μετανάστες και όσο χρόνο χρειαστεί να γίνονται οι Ολομέλειες στις Βρυξέλλες. Ιδού αγαπητοί συνάδελφοι ένα συγκεκριμένο μέτρο που θα επέτρεπε στο κοινοβούλιο μας να συμμετάσχει και αυτό στην προσπάθεια και να δείξει στην πράξη ότι σέβεται τις αρχές της αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης. Σας ευχαριστώ για την ομάδα ευθυντή. Ο κύριος Φάραντς έχει τον λόγο. Κάνατε λάθος πάλι κύριε Γιονκέρ. Σας είχα πει τον Απρίλιο ότι η πολιτική σας για τη μετανάστευση στην ουσία προβλέπει ότι όποιος βάλει το πόδι του στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μείνει για πάντα και δυστυχώς έχουμε αυτή τη στιγμή ένα βιβλικό διαστάσεων μεταναστευτικό κύμα. Ε, στην ουσία οποιοδήποτε μπορεί να έλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα για να φτιάξει κανείς ένα κατάλογο χωρών από τις οποίες κάποιος μπορεί να μείνει ή κάποιος ε, δεν μπορεί να μείνει. Θα λένε όλοι ότι έρχονται από τη Συρία, θα έχουν ένα πλαστό διαβατήριο. Η πλειοψηφία αυτών οι οποίοι έρχονται είναι η οικονομική μετανάστευση. Ε, τολμήστε να το πείτε. Και είναι σαφές πλέον έχουμε δείγματα ότι το ISIS έχει χρησιμοποιήσει αυτό το μεταναστευτικό κύμα για να βάλει πόδι στην Ευρώπη. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε τρελοί να αρνηθούμε την πραγματικότητα. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους πραγματικούς πρόσφυγες, εφόσον θέλουμε να προστατεύσουμε τις κοινωνίες μας και εφόσον θέλουμε εμείς να σταματήσουμε την εγκληματική εκμετάλλευση των ανθρώπων αυτών, πρέπει να σταματήσουμε τα πλοία που έρχονται εδώ, τα σκάφη που έρχονται εδώ και μετά να μιλήσουμε για το καθεστώς της χορήγησης αφήσου. Άκουσα τα σχόλιά σας και για το Ηνωμένο Βασίλειο, για την επίσκεψή σας εκεί. Ε, ξέρω ότι ε, ε, θα ξοδέψετε πάρα πολλά δισεκατομμύρια των Βρετανών φορολογουμένων για να μας πείτε το τι πρέπει να κάνουμε. Θα σας καλωσορίσουμε. Αλλά το να λέτε ότι μειώνοντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία θα μας κάνετε να αλλάξετε, θα αλλάξουμε γνώμη, όχι βέβαια, εφόσον δεν δώσετε τη δυνατότητα στον Κάμερο να ελέγξει τα εξωτερικά του σύνορα για μια ακόμη φορά, mm. τότε δεν θα έχετε πετύχει τίποτα και θα είναι πια πολύ αργά για σας. ENF, e e ο κύριος Φίλιππο έχει το λόγο. Είναι απλό να πει κανείς τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Κρίση, οικονομική κρίση, διπλωματική κρίση. Βλέπουμε τι κάνει το ΝΑΤΟ ή τι θα ήθελε να κάνει στην Ουκρανία, στη Συρία, για όλες αυτές τις χώρες που έχετε καταστρέψει. Και τώρα φυσικά πλημμυρίσαμε από ε, παράνομους μετανάστες. Ανησυχώ λοιπόν και αυτά τα οποία είπατε με κάνουν να ανησυχώ ακόμα περισσότερο. Τα βρίσκω παρανοϊκά θα απευθύνεται 160.000 παρανόμους στα διάφορα κράτη-μέλη ήδη από την επόμενη εβδομάδα και απειλείται με οικονομικά μέτρα τις χώρες οι οποίες θα διστάσουν να το κάνουν αυτό. Οι λαοί της Ευρώπης δεν θέλουν αυτά που ζητάτε πια. Δεν θέλουμε άλλα προβλήματα οικονομικά. Δεν πιέζεται σε καμία περίπτωση όλες αυτές ε, τις μοναρχίες που βασίζονται στο πετρέλαιο. Και ε, σχετικά με τους γεωργούς, δεν τους εκτιμάτε βέβαια. 500 εκατομμύρια τους δίδεται, ενώ δίδεται στους παράνομους μετανάστες 4 δις. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια κρίση. Εσείς προσπαθείτε με το τέρας που έχετε δημιουργήσει να κυριαρχήσετε στον κόσμο. Φωνάζετε ναι στην Ευρώπη. Λες και το πρόβλημα θα λύσει από μόνο του το πρόβλημα και αυτή η υποτιθέμενη ομιλία σας για την κατάσταση της Ευρώπης, της Ένωσης είναι μια αποτυχία. Μέσα από την δημοκρατία, μέσα από τα δημοψηφίσματα, μέσα από την αλλαγή των Βρετανών, τότε θα διαλυθεί το κατασκευασμά σας και θα γυρίσουμε στην ειρήνη και την πραγματική δημοκρατία. Για τους ε, μη εγγεγραμμένους ε, ο μη εγγεγραμμένο βουλευτή, ο κύριος Μορβάη. Κυρία Μορβάη. Patriots unite. Ευχαριστώ. Πατριώτες, ενωθείτε. Πρώτα απ' όλα ήθελα να, πρώτα ήθελα να γράψω Ούγγροι πατριώτες ενωθείτε γιατί ενισχώ για την πατρίδα μου. Μετά ήθελα να γράψω πατριώτε τη Ευρώπη ενωθείτε. Γιατί γνωρίζω πως πολλοί πατριώτες στην Ευρώπη αισθάνονται το ίδιο. Και τέλος συνειδητοποίησα πως υπάρχουν πατριώτες όχι μόνο στις χώρες προορισμού και διέλευσης αλλά και στις χώρες προέλευσης, στις αφρικανικές χώρες, στις φτωχές χώρες της Ασίας. Όλοι έχουμε το ίδιο όνειρο. Να ζούμε στην πατρίδα μας. Να δουλεύουμε στην πατρίδα μας με ειρήνη. Να κρατήσουμε τις ρίζες μας, τον πολιτισμό μας, τις παραδόσεις μας. Να ενωμένοι και ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να εργαζόμαστε για το κοινό μας όνειρο και ας γίνει ο κόσμος ένα καλύτερο μέρος. Σας ευχαριστώ. Im Namen des äh, Rates Κύριε Πρόεδρε, και κύριοι, αγαπητά μέλη, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Επίτροπε, εξ ονόματος του Συμβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Γιούνκερ για την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, για την ε, εξαιρετική ανάλυση που έκανε της κατάστασης σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ονομάτισε τα πράγματα και κυρίως γιατί έκανε προτάσεις. Έκανε προτάσεις σημαντικές και αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες. Έχετε δίκιο κύριε Πρόεδρε όταν λέτε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μιλάμε για business as usual. Τώρα απαιτούνται δράσεις, θαραλέες και καινοτόμες εξαιρετικές δράσεις οι οποίες να κινητοποιούν το δυναμικό της Ένωσης. Εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Έχουμε μια ιστορική στιγμή, βιώνουμε μια ιστορική στιγμή μπροστά μας και το ίδιο έγινε και την εποχή της πτώσης του τείχους και της επανένωσης της Υπήρου μας. Η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει μια μεγάλη κρίση. Απαιτείται αλληλεγγύη, απαιτείται ε, ε, ενέργεια και θάρρος. Ο πρόεδρος Γιούνκερ επέμεινε στα θέματα της μετανάστευσης και στα θέματα των προσφύγων. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πρόσφατα γεγονότα μας το επιβεβαιούν. Έχουν ε, αρχίσει να παίρνουν διαστάσεις τις οποίες δεν υποπτευόμεθα στο παρελθόν. Έχουν αρχίσει να μας ξεπερνούν έχουν αρχίσει να αμφισβητούν τις αξίες μας, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και τους κανόνες μας. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να κολλησιεργούμε, δεν μπορούμε να καθυστερούμε χωρίς λόγο. Ε, στο Συμβούλιο Τζάι του μηνός Ιουλίου η Προεδρία συγκέντρωσε την προσοχή της έτσι ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ειδικά με τον προσωρινό έκτακτο μηχανισμό επανεγκατάστασης ε, των προσφύγων. Δεν σας κρύβω ότι η προσπάθεια αυτή δεν ήταν διόλου εύκολη. Η προσπάθεια αυτή δεν ήταν και επαρκής. Πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και με υψηλότερες ταχύτητες. Οι προτάσεις τις οποίες έκανε ο κ. Γιούν και σήμερα είναι μια σημαντική συνεισφορά στην τρέχουσα διαδικασία και προβλέπονται νέες συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι τον κατεπήγοντα χαρακτήρα επανένωσης των δυνάμεών μας. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με διαιρέσεις. Είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή. Μιλάμε για το 0,11% του πληθυσμού. Δεν είναι τεράστιοι οι αριθμοί. Αλλά θα το πετύχουμε αυτό μόνο αν δράσουμε σύμφωνα με τις αξίες μας, αποφύγουμε τις εθνικές αναδιπλώσεις και εφαρμόσουμε μια ουσιαστική κοινή πολιτική. Η Προεδρία κάνει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε συνεργαζόμενοι με όλα τα κράτη-μέλη και σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα μεταξύ των οποίων και το δικό σας. Αυτό απαιτεί προσπάθειες, προσπάθειες από όλους και θα επανέλθω σε αυτά στην συζήτηση η οποία θα γίνει ειδικότερα για τα θέματα της μετανάστευσης. Κύριε Πρόεδρε, είχαμε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε και τις ε, υπόλοιπες προτεραιότητες της Προεδρίας μας οι οποίε συμπίπτουν εν με αυτές τις οποίες προανέφερε ο Πρόεδρος τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ανεργία, η ανάκαμψη η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί και να ενθαρρυνθεί, τα προβλήματα της ανεργίας των νέων. Έχουμε ένα πρόγραμμα επενδύσεων το οποίο θα πρέπει με θάρρος και με ταχύτητα να θέσουμε σε εφαρμογή. Η Λουξεμβουργιανή Προεδρία υπολογίζει πολύ σε εσάς και νομίζω ότι συμβαδίζουμε εδώ, είμαστε στο ίδιο μήκος κείμενο, Κείμαστε τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε την κοινωνική διάσταση και παρατήρησα αυτά τα οποία είπατε για το κοινωνικό ντάμπινγκ και για την εφαρμογή της αρχής ίδια εργασία, ίδια αμοιβή. Πρέπει να διατηρήσουμε τα κοινωνικά κεκτημένα, Πρέπει να δημιουργήσουμε μια σωστή ισορροπία από τη μία ανάμεσα στα κοινωνικά δικαιώματα και από την άλλη στην ελευθερία την οικονομική. Πρέπει να στηρίξουμε την εσωτερική αγορά ιδιαίτερα στον τομέα του ψηφιακού κόσμου. Μετασχηματίσει όχι μόνο τη βιομηχανία μας και τις υπηρεσίες, αλλά και τον τρόπο που εργαζόμαστε. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι αλλαγές θα υπάρξουν στην αγορά εργασίας, τι επιπτώσεις θα υπάρξουν στο θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης. Οι μεγάλες προκλήσεις της αηφόρου ανάπτυξης, η καταπολέμηση της υπερθέρμανσης απαιτούν την κινητοποίηση των προσπάθειών μας πριν από τη συνάντηση στο Παρίσι. Και η COP21 είναι ένα σημαντικό ραντεβού γιατί η πρόκληση είναι σημαντική. Να μην ξεχνάμε ότι αυτή η κρίση των προσφύγων είναι εν πολλής το αποτέλεσμα άλλου είδους κρίσεων, άλλων σειράξεων στην ευρωπαϊκή γειτονία. Και όταν βλέπω το τι συμβαίνει, δεν θα έλεγε και κανείς ότι η γειτονία μας αυτή είναι ιδιαίτερα σταθεροποιημένη. Διασχίζεται από συνεχείς συγκρούσεις και σειράξεις. Η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να είναι ένας διεθνής εταίρος με θεμελιώδη ρόλο, με την προσπάθεια της Φεντερίκα Μογκερίνη. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς και η διεθνής κοινότητα να αναλάβουμε δράση και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Σας ευχαριστώ κύριε Σμιτ. Για την ομάδα του ΕΛΚΟ κύριο Ρόιλ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής του Συμβουλίου του Κοινοβουλίου. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον ε, κύριο Γιούνκερ που ξεκαθάρισε πως ε, η Ευρώπη είναι κάτι ευρύτερο από τα οικονομικά, ότι είναι και θέμα αξιών και ίσως το ζήτημα των προσφύγων είναι μια ευκαιρία να επανέλθουν αυτά τα ζητήματα στο κέντρο. Υπάρχει, υπάρχουν θέματα ιστορίας, ε, συμβάσεων, αξιών. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε και λογικό είναι πράγματι τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτό που τους αναλογεί και σωστά αναφέρθηκε πως υπάρχει μια δεύτερη πτυχή. Δηλαδή, ασφαλείς χώρες προέλευσης να οργανωθούν οι επαναπατρισμοί, να καταπολύσουμε τους διακινητές. Δεν είναι απλό το ζήτημα να βρούμε μια μαγική λύση όπως ε, θεωρείται ότι είναι παραδείγματο χάρη η νόμιμη ε, μετανάστευση και μόνο έτσι το λύσαμε. Εδώ όμως δεν άκουσα το εξής πάρα πολύ απλό. Πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά και πώς θα ακολουθήσουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Γιατί αυτό θα γίνει μόνο εάν οι ε, Ευρωπαίοι πολίτες έχουν ευημερία και πλήρη ανάπτυξη και αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο στην Ελλάδα. Οπότε θα πρέπει να βρούμε μια ευκαιρία να σκεφτούμε πώς θα υπάρξει ανάπτυξη στην Ευρώπη. Τι γίνεται με την εσωτερική αγορά, τι γίνεται με τους ε, κανόνες μας τι γίνεται με τις τιμές ε, της ενέργειας, με την καινοτομία και την έρευνα. Αυτά ως ερωτήματα, γιατί δεν μου έχετε δώσει και περισσότερο χρόνο, αλλά αυτά είναι προϋποθέσεις για να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Monsieur le Κύριε Πρόεδρε, ο λόγος σας ήταν θαραλέος υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης των Ευρωπαίων και σας υποστηρίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή κρίση και τελικά το θέμα είναι ότι πρέπει να αναρωτηθούμε τι άνθρωποι είμαστε εμείς οι Ευρωπαίοι. Σε τέτοιες κρίσεις, τέτοιες κρίσεις μπορούν να λυθούν μόνο από πραγματικές ευρωπαϊκές προσπάθειες. Αυτή η τραγωδία που βλέπουμε μπροστά μας και στα σύνορά μας, η ανθρωπιστική κρίση που έχει ξεφύγει τελείως, σημαίνει ότι η μόνη λύση είναι ένα πραγματικό σύστημα ευρωπαϊκού ασύλου, ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Η μόνη λύση, επαναλαμβάνω, είναι πραγματική, πραγματικό ευρωπαϊκό πρόβλημα για τη μετανάστευση και αναπτυξιακή συνεργασία. Αυτές τις εντάσεις που βλέπουμε στην αγορά εργασίας η μόνη λύση είναι να επιστρέψουμε όπως είπατε και εσείς σε ένα πρόγραμμα για πλήρη απασχόληση στην Ευρώπη και το επενδυτικό σχέδιο είναι το κύριο εργαλείο γι' αυτό. Μπορούμε όμως να πούμε ότι όλες οι χώρες μέλη έχουν συνθήκες, τις ικανές ε, συνθήκες εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω εφόσον η Ευρωζώνη είναι χώρος διαφοράς και όχι σύγκλησης. Γι' αυτό το σχέδιό σας για τη συμπλήρωση της ΩΝΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Για να καταλήξω λοιπόν Πράγματι χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή λύση και γι' αυτό εμείς οι κοινοβουλευτικοί πρέπει να εκπροσωπήσουμε όχι μόνο τους πολίτες των χωρών μας, αλλά τους Ευρωπαίους πολίτες συνολικά. Τελεία. Ευχαριστώ. Δεν θα δώσω μπλε κάρτα γιατί έχουμε καθυστερήσει και παρακαλώ όλους τους ομιλητές να σέβονται αυστηρά το χρόνο τους γιατί μετά θα γίνουν και ψηφοφορίε και έχουμε και άλλε συζητήσει το απόγευμα και γι' αυτό θα είμαι υποχρεωμένο αντίθετα από ό,τι συνέβαινε πριν να είμαι αυστηρότατο για το ωράριο και το χρόνο ομιλία. Κύριος Τελικάμπρας. Κύριε Γιόνκερ, ξέρουμε ότι η κατάσταση αυτών των προσφύγων που καταφέρνουν να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια είναι καταστροφική. Τεχνικές και πολιτικές λύσεις χρειαζόμαστε επιγόντως. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι. Αναφερθήκατε στις ρίζες του προβλήματος. Ωραία, εγώ θα ήθελα να ε, μιλήσω για την ηθική διάσταση του προβλήματος που φαίνεται να αποφεύγουν όλοι. Το Συμβούλιο, και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο οφείλουν να αναγνωρίσουν, να αναγνωρίσουν ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες σε μεγάλο βαθμό, όχι αποκλειστικά, αλλά σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνε για την τωρινή κατάσταση. Όχι μόνο για την ε, εισβολή στο Ιράκ, στο παρελθόν, αλλά διότι ευθύνονται για τη συμμετοχή τους σε πολλές ένοπλες σειράξεις στη Μέση Ανατολή και στη Μεσόγειο γενικότερα που μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Από πλευράς ήθους και δικαιοσύνης αυτό θα έπρεπε να το αναγνωρίσουμε. Και αυτό θα διευκολύνει και την ανάληψη άλλων βημάτων που τόσο χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Καστάλντο. Ευχαριστώ. Μας μιλήσατε για την καθοριστική στιγμή στην οποία έχουμε βρεθεί σήμερα. Ο κύριος Τούσκ ε, απουσιάζει. Είναι λυπηρό, διότι θα έπρεπε να μιλήσουμε για την κατάσταση της Ένωσης, αλλά για τις καταστάσεις και τα κράτη της Ένωσης. Ε, να μιλάμε για το Μαρενόστρουμ, για το κόστος ε, της μετανάστευσης, Ξεχνούν οι ανατολικές χώρες, οι χώρες Ανατολικής Ευρώπης, την περίοδο που ε, οι δικοί τους οι πολίτες ήταν πρόσφυγες. Ξεχνούμε οι πολυεθνικές μας τι κάνουν στον κόσμο και σε ποια κατάσταση οδηγούμαστε λόγω αυτής της δράσης τους. Ε, για να μην αρχίσω να μιλάω για την Κίνα και την TTIP και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο Λίβανο, στην ε, η Ορδανία δεν έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες ε, για να ε, δώσουν μια βοήθεια στα αδέλφια τους που βρίσκονται σε αυτή την επικίνδυνη κατάσταση. Το χάσμα διευρύνεται όλο ένα και περισσότερα ανάμεσα στους ισχυρούς και στους ασθενείς. Είναι δειλή η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο δρά, οι αξίες ε, που πρεσβεύει θα έπρεπε να είναι εφαρμοστές για όλους, για τους συμπολίτε μας, αλλά και για τους μετανάστες και πρόσφυγες. Ας μην επιλέγουμε την οδό της ευκολίας. Ε, μόνο με τη δικαιοσύνη θα αποκαταστήσουμε την ειρήνη. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δεγκράφ, σας παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο αγόρευσης, ε, γιατί έχουμε, έχουν σημειωθεί υπερβάσεις ήδη από τους συναδέλφους σας. Πρόεδρε, σήμερα ο πρόεδρο Γιούγκερ μα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα για να υποδεχτούμε 160.000 μετανάστε στην Ευρώπη. Δεν είναι το σχέδιο Γιούγκερ αυτό, είναι το σχέδιο Μέρκελ, α το πούμε έξω από τα δόντια ε, που θέλει να επιβάλλει η κυρία Μέρκελ και ο πρόεδρο ο, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι η δημοκρατία λοιπόν στην πράξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία βλέπει ότι δεν μπορεί να υποδεχτεί όλο τον κόσμο και αφήνει τον υπόλοιπη Ευρώπη να λουστεί όλα όσα έκανε αυτή και να δώσει δωρεάν χρήματα στους έτοντες άσελου. Δεν ε, λέει αυτό το πρόγραμμα, αυτό ότι θα σταματήσουμε να δίνουμε δωρεάν χρήματα. Και αυτό το πρόγραμμα συνδέεται με το Σέγγεν περά το γεγονός ότι μέσα, ανάμεσα στους ε, πρόσφυγες υπάρχουν πολλοί και τρομοκράτες και μέλη της ο κύριος Γιούνκερ λοιπόν θα πρέπει να πάει στην κυρία Μέρκελ και να της τα ξαναεξηγήσει. Να δείξει αλληλεγγύη με τον Ευρωπαίο πολίτη, με την ασφάλειά του, να κλείσει τα εθνικά σύνορα και να σταματήσει να δίνει για εκατοντάδες χιλιάδες τεχοδιώκτες ε, δωρεάν ε, χρήματα, ενώ τόσοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν στην φτώχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Όλμπρεχτ. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, εξ ονόματος της Πολωνικής ε, Αντιπροσωπεία και του ε, Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εκφράζουμε ότι συμπάσχουμε, κύριε Γιούγκερ. Ε, Εξέλισσεται κι άλλο η κατάσταση και θα ήθελα εξ ονόματος της Πολωνικής Αντιπροσωπείας να πω το εξή, γιατί όλοι από μια χώρα είμαστε. Εμείς είμαστε από μια χώρα η οποία έχει ανατολικά σύνορα, ανατολικά σύνορα Είπατε ότι η κατάσταση, και δικαίω είπατε, ότι η κατάσταση με την Ουκρανία μπορεί να επιδεινωθεί δραματικά. Είναι πάρα πολύ ε, ευάλωτη η κατάσταση. Δεν ξέρουμε πώ μπορεί να εξελιχθεί. Και πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται μόνο ανακατανομή, ότι χρειάζεται μια δυναμική αντίδραση για το πρόβλημα αυτό. Είναι τόσο τραγική η κατάσταση που στην Πολωνία φυσικά και αντιλαμβανόμαστε την ανθρωπιστικό δράμα, αλλά καλούμαστε να συζητήσουμε το κατά πόσον μπορούμε καν να υποδεχθούμε πιο πολλούς πρόσφυγες. Έχουμε μια τέτοια πρόταση επιτάπητος, αλλά θεωρούμε ότι ο έλεγχος για τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να παραμείνει στα εθνικά χέρια. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κάτι ακόμα. Είμαστε από χώρε όπου γνωρίζουμε πολύ, ακριβό, πολύ καλά ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αλλά δεν θέλουμε να επιτρέψουμε να μας ε, εκδιάζουν με ευρωπαϊκούς πόρους, να μας ασκήσουν πίεση. Είμαστε λοιπόν υπέρ μιας λύσης, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει Σαλόμ. Όταν, ε, πρόεδρε, θέσουμε ένα τέρμα ε, σε αυτή τη ε, διαδικασία που τώρα ξεκινάει, θα έχουμε φτάσει ήδη στο ίμιση της θητείας μας. Και θα έλεγα ότι οπισθοχωρούμε από κοινωνικής πλευράς τουλάχιστον μία δεκαετία με αυτά που συμβαίνουν τώρα. Θα έπρεπε να το αποφύγουμε πάση θυσία. Δηλαδή η έξοδος από την κρίση δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι θα θυσιάσουμε τα κοινωνικά μας κεκτημένα. Θα πρέπει να προασπίσουμε τα κοινωνικά μας δικαιώματα, να καταπολεμήσουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ. Για την ανθρωπιστική κρίση Αυτά τα 160 εκατομμύρια εκτοπισμένων ανθρώπων προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, από την πείνα και σήμερα υπάρχουν ε, περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο που πεθαίνουν από την πείνα από αυτούς που πεθαίνουν ε, λόγω ενόπλων σειράξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάσκεψη που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη την ερχόμενη άνοιξη θα πρέπει να περάσει ένα ηχηρό μήνυμα για να μείνουμε εξάλλου και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου το Δεκέμβρη. Στην Κωνσταντινούπολη θα έπρεπε ιδανικά να αποδείξουμε αυτά που έχουμε ήδη καταφέρει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αλλά αν δεν δείξουμε αλληλεγγύη δεν θα μπορέσουμε να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο στην Κωνσταντινούπολη. Ο κύριος Λόντγκριν, ευχαριστώ. Τι, έχω ένα λεπτάκι στη διάθεσή μου και θα ήθελα να συζητήσω την κατάσταση στην ε, Ουκρανία, γιατί αναφέρθηκε και ο κύριος Γιούγκερ. Από ρωσικής πλευράς, αυτά που γίνονται στην Ουκρανία δεν είναι κάτι που μπορεί να θεωρηθεί αξιοπρεπές ε, ε, με τα μοντέρνα δεδομένα πρόκειται για βία, για διωγμό νέος ολόκληρου λαού στην Ουκρανία και έχουμε ζητήσει ε, από πλευρά της πολιτικής μου ομάδα, όχι μόνο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στο Κοινοβούλιο στη Σουηδία, η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει στις ε, διπλωματικές διαπραγματεύσεις ε, και να αναλάβει αποφασιστικότερα τη δράση. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε την Κρυμαία και την Ουκρανία στα χέρια της ε, Ρωσίας. Ε, πρέπει να δράσουμε τώρα. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγους μήνες ε, μας απείλησε η Ρωσία ότι θα σταματήσει και την παροχή του αερίου. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του Ουκρανικού λαού. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε την απαιτούμενη δράση για να επιληθεί επιτέλους αυτή η κρίση και δεν αντέχει άλλο ο λαός της Ουκρανίας. Ευχαριστούμε κύριο Άκτινσον. Ο Λαμασούρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το όραμα, τον ηγετικό ρόλο που επιδεικνύει το ευρωπαϊκό του πνεύμα ε, όλες αυτές οι ιδιότητες ε, δυστυχώς ε, σε πολλές περιπτώσεις λείπουν από τον πολιτικό βίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέτε ότι δεν πρέπει να κρύβουμε την ομοία αλήθεια και συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχει μια έλλειψη ένωσης μέσα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν λειτουργεί εύρεθμα όπως θα έπρεπε. Η πολιτική μας τίθεται στο βωμό των εθνικών συμφερόντων. Δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τι υποχρεώνεται να αποφασίζει με ομοφωνία ε, σε εθνικιστικά συμφέροντα εκεί όπου θα έπρεπε να επικρατεί το κοινό καλό. Κάνει ε, συζητήσεις για κλεισμό των θυρών ε, για τη μετανάστευση τον Ιούνιο έγιναν αναξιοπρεπή επέσχυντα, επέσχυντες διαπραγματεύσεις και επιλέγονται κοντόφθαλμες λύσεις εις βάρος μακροχρόνιων πολιτικών. Το Συμβούλιο μέσω της αμέλειας του, μέσω της υποκρισίας του, τι έχει κάνει αφήνει τους Υπουργούς Οικονομικών που τώρα εξετάζουν το σχέδιο προϋπολογισμού το 2016 να περικόψουν όλες τις γραμμές που χρησιμεύουν για να χρηματοδοτηθεί η πολιτική μετανάστευσης και ασύλου. Ήρθε η ώρα ε, να επικρατήσει μεγαλύτερη ομοθυμία μέσα στην Ένωση. Ε, ευχαριστώ κύριο Βένταν Όλσεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Γιούγκ, ε, θα ήθελα με κάθε ειλικρίνεια να σας ευχαριστήσω γιατί πραγματικά έχει έρθει η στιγμή της αλήθειας και έχει έρθει η στιγμή και για περισσότερη Ευρώπη. Το θέμα των προσφύγων θα καταστεί η λιδία λίθος για τους Ευρωπαίους. Αν δεν τα καταφέρουμε μπορεί να χάσουμε τα πάντα αλλά μπορεί και, μπορεί και να κερδίσουμε πάρα πολλά. Σας είμαι λοιπόν ευγνώμων που δεν συρρυκνώσατε τη συζήτηση μόνο στο θέμα των ποσοστώσεων ε, που ε, αναφερθήκατε στη συνεισφορά συμπεριφορά των κρατών της Μέσης Ανατολής και για να είμαι ειλικρινής για αυτές τις χώρες προσφέρουμε πάρα πολλά, πολύ λίγα. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία και δεν αρκεί να παραπέμπει κανείς στα hot spot που θα διατίθενται. Αυτή τη στιγμή ε, στα Βαλκάνια δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι καθοδόν, ε, ζουν στην Ήπετρο όταν βρέχει όπω βρέχει σήμερα. Για του ανθρώπου αυτού μπορεί να προκύψουν ε, αντισόπιες καταστροφές. Παρακαλώ λοιπόν να δραστηριοποιηθείτε και θα ήθελα να στηρίξετε χώρες όπως ε, τη Σερβία η οποία ανέλαβε ένα καθήκον και το εκπληρεί παραδειγματικά. Ευχαριστούμε πολύ ο κ. Γκονζάλες Πόμς. Ο κύριος Γιούνκα ανέφερε ένα παράδειγμα. Η Ισπανία έχει πάνω από 4 εκατομμύρια ανέργους και παρόλα αυτά την ε, πρόταση των, ε, της Κομισιόν τους πρόσφυγες θα την υιοθετήσουμε και για λόγους ανθρωπιστικούς αλλά και γιατί ως Ευρωπαίοι νιώθουμε ότι έχουμε αυτό το καθήκον. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το φανατισμό και τον πόλεμο. Ο κύριος Γιούγκα ανέφερε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τους δικούς μας τους πολέμους ε, και τη δυστυχία που προέκυψε στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μια κοινή πολιτική ασύλου αλλά και μια κοινή πολιτική για εξωτερική ειρήνη. Χρειαζόμαστε χρειαζόμαστε μια πολιτική συμβίωσης, ε, πολιτική ανεκτικότητας, τα σύνορα ε, να καταργηθούν στις καρδιές μας ε, καταρχήν. Αυτή η τραγική εικόνα με το Σύριο παιδί που πέθανε, που έχασε τη ζωή του σε μία ακτή της Τουρκίας ε, συγκίνησε πάρα πολλούς, αλλά δεν είναι το πρώτο παιδί που πεθαίνει. Δυστυχώς έχουν πεθάνει πάρα πολλά πριν από αυτό και θα πεθάνουν και άλλα τόσα. Η Συρία δεν είναι ο μόνος πόλεμος που μένεται στη γειτονιά μας. Θα υπάρξουν ε, κατοντάδες προσφύγων, πρόσφυγες ε, για λόγους κλιματικής αλλαγής, ασθενειών. Η ανακατανομή λοιπόν αυτών των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι δύσκολη Πρόκειται για ένα δύσκολο, ακαθόδη δρόμο και ως εκ τούτου ας μην ξεχνάμε ότι για τα επόμενα έτη θα αντιμετωπίζουμε προκλήσεις. Προκλήσεις που θα μας συνοδεύουν. Τίθεται λοιπόν το εξής ερώτημα. Πόσοι και πότε. Πότε η διεθνής κοινότητα θα οδηγήσει σε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο. Όσο μένεται αυτός ο πόλεμος δεν θα αρκούν ποτέ ποσοστώσεις για να δεχθούμε αυτούς τους ανθρώπους. Η κυρία Περβάνς Περές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως και άλλοι, θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου. Την σημερινή σας ομιλία, που θα έλεγα ότι επανέρχεται στην καρδιά όχι των κοινοτικών μεθόδων αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αξιών της, της αλληλεγγύης της, χωρίς την οποία τίποτα δεν είναι πλέον εφικτό, στην αλληλεγγύη που είναι ε, ο ακρογωνίος λίθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια αξία ε, ιδιαίτερα προσφυλή στη δική μας πολιτική οικογένεια και χρειάζεστε σε μεγάλο βαθμό αυτή την αλληλεγγύη για να μπορέσετε να υλοποιήσετε το θεματολόγιο που μας ε, παρουσιάσατε σήμερα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εμπόδισε το Brexit, γιατί αυτό θα ισοδυναμούσε με ε, κατάλυση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Όμως ε, πρέπει να κάνουμε και άλλες υπερβάσεις. Ε, θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να πραγματευτούμε και το θέμα του χρέους, διότι όλοι ξέρουν ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος, οπότε ας το προσεγγίσουμε με αποφασιστικότητα και με αλληλεγγύη. Και ούτω τρόπος εκφράσατε και την αποφασιστικότητά σας ε, να δείξετε την οικονομική διακυβέρνηση σε ένα εργαλείο που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις, ακόμη και τις προκλήσεις με τις οποίες ε, είναι αντιμέτωπε τα κράτη-μέλη για το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα. Σας ε, παρακαλώ όμως ας μην έχετε μόνο το εργαλείο των κυρώσεων αλλά και των κινήτρων. Χρειαζόμαστε αυτό το καρότο για να μπορέσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βασιστούμε στι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να επιτύχουμε αυτά που θέλουμε. Διακόπτει την κυρία Μπερέσο, ο Πρόεδρος. Ε, Γκαρντίνη παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα για άλλη μια φορά να επιβεβαιώσω ότι είμαστε πολύ υπερήφανοι που μπορέσαμε να στηρίξουμε εσάς, ε, κύριε Γιούγκερ, ε, πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν σας ακούμε να μιλάτε, ε, νιώθουμε ότι ταυτιζόμαστε με αυτά που λέτε γιατί βρισκόμαστε στην ίδια Ευρώπη για την οποία είσαστε πεπισμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ολοκληρωμένη ανθρώπινη αλληλέγγυα παρέμβαση που κάνατε εδώ στην, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Μιλήσατε για τη χριστιανική Ευρώπη και για πάρα πολλά άλλα και αναφέρατε ότι από τη μία πλευρά είναι αλήθεια ότι θα πρέπει σήμερα να ξεπεράσουμε τα εμπόδια, να απαντήσουμε δημιουργήσουμε αλληλέγγυα στην έκτακτη αυτή ανάγκη, να διαθέσουμε τα μέσο μακροπρόθεσμα μέτρα για να μπορούμε να προλάβουμε αυτές τις ε, τραγικές καταστάσεις. Αυτό είναι θέμα καταρχήν ανθρωπιάς και δεύτερον ιστορικής δικαιοσύνης. Ε, εμείς ε, ως Ιταλοί, ως πολιτική ομάδα Φόρτσα Ιταλία μέσα στο ΕΛΚ θεωρούμε ότι πράγματι ταυτιζόμαστε με όλες τις δικές σας προτάσεις και ελπίζουμε το μήνυμά σας να φτάσει ολοκληρωμένο. Γιατί πάρα πολλοί μας παρακολουθούν σήμερα και αυτά που λέμε δεν πρέπει να προκαλέσουν αυταπάτες. Ε, πρέπει να απαντήσουμε στην έκτακτη ανάγκη με λογική, να είμαστε χρήσιμοι για να αποφύγουμε και άλλα δράματα και τραγωδίες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσέγγισή σας. Σας ευχόμαστε ευόντως των εργασιών. Θα σας στηρίξουμε. Η κυρία Τόγια. Πρόεδρε, Είπατε ότι για την Ευρώπη οι στιγμές είναι μοναδικές, εξαιρετικές, ιστορικές. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ισχυρή ε, συλλογική ηγεσία. Το να είναι κανείς ηγέτης δεν μπορεί κανείς να το μάθει, δεν αποκτά πτυχίο ηγέτη. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα ηγέτη που να αναλάβει τα καθήκοντα τα οποία προκύπτουν σήμερα από την Ευρώπη. Σχεδόν δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα την εσωτερική μας κρίση, την οικονομική, την ανεργία και παρόλα αυτά η Ευρώπη πλήττεται από αστάθεια, από κρίση ανθρωπιάς. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητάμε κατηγορηματικά να δείξετε ηγετικό πνεύμα, να δείξετε μια ευρωπαϊκή οδό η οποία θα ξεπερνάει τα εθνικά συμφέροντα. Δυστυχώς μερικά κράτη εξακολουθούν να επιδεικνύουν εγωισμό. Ίσως να είναι οι ίδιες αυτές χώρες οι οποίες όμως ξεχνάνε ότι βρέθηκαν εδώ λόγω της ελεγγύης που τους επιδείξαμε πριν από κάποια χρόνια. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο πρόεδρός μας, ο κύριος Πιτέλα, οι προτάσεις σας να είναι επίκαιρες, κατάλληλες, γιατί δεν μπορεί κανείς πλέον να μιλάμε απλά για την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη πολλές φορές λέει πολλά, αλλά ε, αντιδρά και δρά εκ των υστέρων. Η κυρία Σπυράκη παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν, αυτό ο χειμώνα ξεκινά με την κατάρρευση δύο σημαντικών συλλογικών ψευδεστήσεων. Κατέρευσε δυστυχώς με τραγικό τρόπο η προσήλωση στο δουβλίνο 2 και η ψευδαίσθηση ότι οι χώρε εισόδου στην ευρωπαϊκή ένωση όπως είναι η ελλάδα και η ιταλία αντέχουν να διαχειριστούν μόνες τους το κύμα των προσφύγων τώρα πρέπει όχι μόνο να αυξήσουμε πολύ περισσότερο από το 1% του κοινοτικού αεπ τη χρηματοδότηση για την ένταξη των προσφύγων αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στον υποχρεωτικό καταμερισμό των ευθυνών. εκεί η κομισιόν έχει λόγο και πρέπει να το παρακολουθεί. την ώρα όμως που υποδεχόμαστε στην ελλάδα γιατί στα ελληνικά νησιά καταλήγουν στην κο και στη λέσβο εκατοντάδες οικογένειες με τα παιδιά στην αγκαλιά γιατί οι έλληνες ξέρουμε από προσφυγιά πρέπει να ξέρουμε και ποιοι είναι εκείνοι που πατούν στο έδαφος μας. ως ευρωπαίοι οφείλουμε να διασφαλίσουμε τα σύνορά μας και οι χώρες υποδοχής πρέπει να ενισχυθούν γι' αυτό. αλλά και στην ελληνική κρίση κύριε πρόεδρε κατέρευσε η ψευδαίσθηση ότι ο λαϊκισμός μπορεί να δώσει λύσεις πλέον στην ελλάδα είμαστε πολλοί που πιστεύουμε ότι η νέα κυβέρνηση πρέπει να έχει ως πρώτη της προτεραιότητα τις μεταρρυθμίσεις. η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές πρέπει να είναι σταθερή και να εγγυηθεί ένα ασφαλές οικονομικό περιβάλλον στο πλαίσιο της συμφωνίας φυσικά και το Grexit δεν θα επιτρέψει το τραπέζι δεν θα επιστρέψει στο τραπέζι και δεν θα το επιτρέψουμε να επιστρέψει. θα τα καταφέρουμε με τη συμβολή της ευρωπαϊκής ένωσης όπως το έκαναν οι ισπανοί οι πορτογάλοι και οι ιρλανδοί. σας ευχαριστώ. Vi prego di rispettare i tempi. Non voglio togliere la parola a nessuno, però non mi costringete. Θα ήθελα παρακαλώ να είσαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το χρόνο, γιατί αν διπλασιάζει το χρόνο που σε διατίθεται, θα αναγκαζώ να μην δώσει το χρόνο σε κάποιου συναδέλφου σα. Ο κύριος, η κυρία Πέρε, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Στη ε, πρωτοσέλιδα τον Ιούνιο του 2015 ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτύχε, απέτυχε για να, την ανακατανομή των προσφύγων και η Ισπανία απέρριψε την ε, κλίδα κατανομής που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εθνικά συμφέροντα και ο εγωισμός αποτελούν το εμπόδιο στο μονοπάτι μας στην αντιμετώπιση της, της κρίσης αυτής που την αντιμετωπίσουμε τα τελευταία χρόνια. Αλλά προφανώς έχουμε και άλλα θέματα και άλλες πτυχές οι οποίες είναι ουσιώδεις. Η Ευρώπη δεν πρόκειται να εξέλθει από την κρίση και να δημιουργήσει ανάπτυξη αν δεν επενδύσουμε και σε άλλους τομείς. Άρα καλωσορίζουμε τα πρώτα βήματα που γίνονται από το σχέδιο Juncker. Αλλά πού είναι η κοινωνική Ευρώπη, πού είναι η καταπολέμηση της ανισότητας, πού είναι οι πρωτοβουλίες που θα εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο μισθό, ένα το μισθό. Και τι γίνεται για την, ε, τις πρωτοβουλίες για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, για την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ. Κύριε Γιούνκερ, ο κερνός περνάει και δεν πρόκειται να περιμένουν την Ευρώπη, ξέρετε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, ο κύριο Κάρα, έχετε επενδύσει πάρα πολύ για την οικοδόμηση μια κοινή συνείδηση. Από πού ερχόμαστε, ποιοι είμαστε και που πού προς τα πού οδεύουμε. Αυτό ήταν και καλό και απαραίτητο η ιδέα της Ευρώπης. Το πολιτικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πολιτικό project αποτελεί το πρόγραμμα εργασίας μας λοιπόν. Ο εθνικός εγωισμός, η ατολμία, η έλλειψη ειλικρίνειας, οι αντιφάσεις μεταξύ των πράξεων και των όσων λέγονται, αυτά αποτελούν το πρόβλημά μας. Και σε εμά εναπόκειται να αλλάξουμε δρόμο και αν αλλάξουμε δρόμο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι. Και σήμερα βλέπουμε πάρα πολλά ε, δείγματα που μας δίνουν τόλμη και θάρρος για την ε, κοινωνία των πολιτών, για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, για τη δημόσια, την συμμετοχή του κοινού. Τα κύματα των προσφύγων, η Ελλάδα, η πείνα, είναι γεγονότα, γεγονότα τα οποία είναι στην πηγή μιας ε, κοινής ε, πρόκλησης της ε, ευρωπαϊκής ε, πολιτικής για την εξωτερική πολιτική, για την άμυνα και για την κοινωνική ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίτερμιουλερ λέει ο Πρόεδρος. Κυρίε και κύριοι, η αλλαγή πάντα αποτέλεσε κινητήρια δύναμη για την Ευρώπη, για να προσαρμοστούμε σε έναν νέο κόσμο. Αυτή η κρίση των προσφύγων ε, σημαίνει το εξή. Είτε θα αλλάξουμε για να ξεπεράσουμε την κατάσταση και θα καταστούμε πιο ισχυροί, ή θα αφήσουμε κατά μέρο τι βασικέ μα αρχέ, τι βασικέ μα αξίε. Και έτσι θα αφήσουμε κατά μέρο και το μέλλον μα. Δεν μπορούμε αυτό να το ε, ανεχτούμε. Έχουμε κακού συμβιβασμού, έχουμε νόμου που είναι παροχημένοι, έχουμε ηγέτε οι οποίε δεν τηρούν τα λόγια του. Δεν μπορούμε να αφήσουμε του πρόσφυγε να κοιμούνται στου σταθμού τρένου και να είναι τα θύματα των διακινητών. Θα πρέπει να αναλάβουμε καινούργιες πρωτοβουλίες, θα πρέπει να υπάρχει κλίτα κατανομής, αλλά αυτό είναι μια αρχή και μόνο έχουμε μεγάλη ευθύνη και δεν έχουμε καθόλου χρόνο να χάσουμε. Θα πρέπει να υπολογίζουμε σε μεγαλύτερη αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη προς ε, τους πρόσφυγες. Σε αυτά βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Δραγγέλ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, κύριε Γιούγκερ, αυτό το θέμα της κρίσης και της μετανάστευσης έχει και ένα πλεονέκτημα για μας τους Ευρωπαίους ε, Μπορούμε να δείξουμε ότι όχι μόνο σε αυτό το τομέα αλλά και σε άλλους ε, χρειαζόμαστε περισσότερη ολοκλήρωση, περισσότερο συντονισμό, περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη. Και γι' αυτό ήθελα να σχολιάσω τώρα το θέμα των ε, δημοσίων οικονομικών που ταλανίζει την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, πολλές άλλες χώρες επίσης ε, που έχουν κάνει απίστευτες θυσίες, κυρίως στα πλαίσια της, στην περίπτωση της Ισπανίας, της Πορτογαλίας,

και της Ιρλανδίας. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξή Ο Πρωθυπουργό μας ήταν ο μόνος που είχε μέχρι στιγμής ένα όραμα για την Ευρώπη. Πρότεινε λοιπόν ο Πρωθυπουργό μας αυτός ο μηχανισμός των ασύμετρων σοκ να μας οδηγήσει σε ένα ε, κοινό ταμείο ανεργίας ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο των τεσσάρων Προέδρων και των έξι Προέδρων 2012 ε, δηλαδή και αυτό που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο μας οδηγήσουν σε ένα τέτοιο μέτρο. Ευχαριστώ τώρα στο Catch the Eye και θα ήθελα παρακαλώ όσοι λάβουν τον λόγο να μην ξεπεράσουν το ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Κίρτσος. Κίρτσος. Αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Γιούνκερ για το θεωρητικό του ρόλο στη διαχείριση της ελληνικής κρίσης. Μετά θέλω να παρατηρήσω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν εντυπωσιακέ πολιτικές εξελίξεις ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει στι εκλογέ με ένα πιο ήπιο πρόγραμμα και η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα μου, κάνει εντυπωσιακά πολιτικά ανοίγματα για συνεργασίε αμέσω μετά τι εκλογέ. Θέλω να τονίσω ότι η πολιτική εξελίσσεται στην Ελλάδα αλλά η οικονομική κρίση παραμένει μαζί μα. εάν αποδείξουμε μετά τι εκλογέ ότι είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε αποτελεσματικά την κρίση θα χρειαστούμε πάλι τη βοήθεια του κυρίου Γιούνκερ και των θεσμών για μια πιο ελαστική πολιτική σε ό,τι αφορά τη φορολογία των αγροτών τη φορολογία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τη φορολογία του τουριστικού τομέα. πρώτα να αποδείξουμε εμείς ότι είμαστε συνεπείς και μετά να χαλαρώσει κάπως η φορολογική πολιτική για να βγούμε από την κρίση με δυναμική οικονομική ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπλάνκο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή θα πρέπει να αντικατροπτίζει και έναν άλλο τομέα που πλήττεται από την κρίση, τους ε, τους ε, αγρότες, οι οποίοι επιθυμούν ε, σωστές τιμές για τα προϊόντα τα οποία παράγουν για το γάλα. Αν δεν υπάρξει άμεση απάντηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν δεν ε, οριστούν κάποιες ελάχιστες τιμές για την παρέμβαση, στην περίπτωση αυτή ο γαλακτοκομικός κλάδος θα καταρρεύσει εντελώς εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις στην καλλικία μεταξύ άλλων. Είναι λοιπόν σημαντικό να ακούσουμε και τους αγρότες που έχουν ξεχυθεί στους δρόμους αναζητούν μία απάντηση. Θα πρέπει να δοθεί μία απάντηση άμεσα. Θα πρέπει να είναι μία δίκαιη απάντηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κινηθεί. Θα πρέπει να ορίσει κάποιες ελάχιστες τιμές παρέμβαση προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπία στην αγορά. Ο κ. Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε την 80 λεπτή ομιλία του κυρίου Γιούνκερ, την οποία ομολογουμένως θα ζήλευε σε διάρκεια ακόμη και ο Φιντέλ Κάστρο μιλώντας για το ελληνικό ζήτημα ο κύριος juncker αναφέρθηκε στη δίθεν προσφορά του προς την ελλάδα τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ πακέτο. Πούλησε δηλαδή για άλλη μια φορά φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Γιατί αυτά τα 35 δις ευρώ είναι κονδύλια που δικαιούται έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014-2020. Ακούσαμε επίσης τον κύριο Γιούνκερ ως κοινικό εκπρόσωπο της Ευρώπης των δανειστών να απειλεί τον ελληνικό λαό αν δεν υποταχθεί στο τρίτο μνημόνιο. Πρέπει λοιπόν κύριε Γιούγκερ να πάψετε να ενεργείτε ως μέλος της Τρόικας. Πρέπει κύριε Γιούγκερ να πάψετε να ενεργείτε ως εκπρόσωπος της νεοαπικιακής γερμανικής Ευρώπης. Σας λέω λοιπόν κύριε Γιούγκερ ότι οι απειλές σας κατά του ελληνικού λαού δεν πρόκειται να περάσουν. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβετε τόσο το καλύτερο για σας και την Κομισιόν. Ευχαριστώ. La parola all'onorevole Pagazzortunava. Ο κύριος Πακατζοτουνάβα. Non è in aula? Από ό,τι φαίνεται όμως δεν είναι στην αίθουσα. Α, είναι η κυρία Πακατζετουνάβα. Κύριε Γιούγκα, Σήμερα σας ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σας, γιατί δείξατε πάρα πολλά ευρωπαϊκά προβλήματα και υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ότι πολύ συχνά ε, πολλοί επικαλούνται την Ευρώπη, αλλά κατ' ουσίαν απλά ε, καταφεύγουν στον εγωισμό τους. Έχουμε σήμερα στην Ευρώπη την κρίση, την κρίση τη μεταναστευτική, την οικονομική. Κάθε κρίση που ακολουθεί είναι και χειρότερη από την προηγούμενη. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε τώρα είναι οι ικανότητε. ικανότητες. Ε, ο εθνικισμός και η αδυναμία μας ε, δεν είναι καλά και θετικά στοιχεία, αλλιώς μπαίνουμε σε ένα τοξικό κύκλο, σε λαϊκισμό. Αυτό οδηγεί σε αντιδημοφιλείς συμπεριφορές, ε, Ουγγαρία, Βρετανία και αλλού. Ε, κύριε Γιούγκα, ε, εσείς μπορείτε να στηρίζεστε στη δική μας την υποστήριξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λόγο έχει τώρα η βουλευτής κυρία Φορέντσα. Κύριε Πρόεδρε, εγώ πιστεύω ότι σήμερα το πρωί είχαμε μια ιστορική σημασία σε συζήτηση. Επιτρέψτε μου να πω ότι ε, διαπίστωσα να υπάρχει εδώ υποκρισία. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει διαφοροποίηση ή ε, η διαφοροποίηση που γίνεται εδώ ανάμεσα σε μετανάστες και πρόσφυγες, οικονομικούς μετανάστες και πρόσφυγες, είναι εικονική. Γιατί εμείς τελικά πρέπει να σώσουμε τους ανθρώπους που θέλουν να ξεφύγουν ε, από τη φτώχεια, από προβλήματα. Όλα αυτά μόνοι μας τα προκαλέσαμε. Πολύ συχνά μιλάμε για μια έκτακτη κατάσταση, μιλάμε για μεταναστευτικές ροές, αλλά κατ' ουσίαν θα έπρεπε να συζητάμε για τη δομική αλλαγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη μεταρρύθμιση του δικαίου περί ασύλου, τη μεταρρύθμιση ε, των διατάξεων περί ευρωπαϊκής υπηκότητας. Οφείλουμε να καταργήσουμε όλους τους ε, τείχους ε, και να μην καταφεύγουμε σε στερεότυπα ότι θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να μείνουν στην πατρίδα τους, στη στιγμή που εμείς οι ίδιοι καταστρέψαμε τα σπίτια τους. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, οφείλω να ομολογήσω ότι σήμερα εντυπωσιάστηκα από ένα μεγάλο κομμάτι της ομιλίας σας. Όχι βέβαια για το TTIP, επ' αυτού ε, εμείς και άλλοι διαφωνούμε. Όμως το μεγαλύτερο κομμάτι της ομιλίας σας, ε, η ελεγγύη για τους ε, πρόσφυγες και για το ότι πρέπει επιτέλους να δραστηριοποιηθούν τα κράτη-μέλη, υποκλίνομαι κύριε Γιούγκα. Θεωρώ βέβαια ότι όλα αυτά τα εννοείται σοβαρά. Είπατε πολύ σωστά ότι είναι αφύσικο να περικόπτει κανείς ε, την αναπτυξιακή βοήθεια. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε τις δυνατότητες να βοηθήσουμε αυτούς που θέλουν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και ελπίζω να το εννοείται και σοβαρά ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι πρόσφυγες θα πρέπει να μπορούν να εργάζονται, να κερδίζουν τα δικά τους χρήματα. Όταν ήσασταν αρχηγός ε, κυβέρνηση, αυτό δεν το θέλετε. Ελπίζω τώρα που το λέτε να το θέλουν άλλοι αρχηγοί κυβερνήσεων. Και θα ευχόμουν να έχουμε εδώ έναν εκπρόσωπο του Συμβουλίου που συμφωνεί μαζί σας και όχι κάποιον ο οποίος και αυτός ε, συμφωνεί με την ανέγερση τείχων. Να έχουμε κάποιον που θέλει αλληλεγγύη στην Ευρώπη όπως και εσείς. Πρόεδρος, Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Λούνατσεκ και τώρα για να ολοκληρωθεί η συζήτηση θα ήθελα να δώσω το λόγο και πάλι στον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Γιούγκερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε πρόεδρε. Ε, μίλησα τόσο πολύ κατόπιν τούτου αυτό που μου ζητήσατε εσείς ως πρόεδρος, να μην μακρηγορήσω στην ε, δεύτερη παρέμβασή μου. Ε, θα το προσπαθήσω. Τώρα κατά πόσο θα τα καταφέρω θα δείξει. Αλλά προφανώς και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να διακόψει τον πρόεδρο της Κομισιόν. Εγώ αν το κάνετε ευχαρίστως ε, θα ε, υποκύψω στην παρέμβασή σας, στην παρένεσή σας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω το εξής. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν εκπροσωπείτε εδώ το Συμβούλιο έχουμε έναν αρμόδιο Λουξεμβούργιο Υπουργό, Υπουργό Εργασίας, ε, ο οποίος ασχολείται εδώ και χρόνια και με την ανάστευση. Αν στο Λουξεμβούργο υπάρχει κάποιος που γνωρίζει τα θέματα, αυτός είναι ο παριστάμενος εκπρόσωπος ε, του Συμβουλίου προεδρεύων ε, αυτό το εξάμεινο. Κατά τα άλλα να πω και το εξής. Κοιτάξτε, δεν είναι σωστό τον ε, κύριο Τούσκ ε, να τον επικρίνει κανείς ε, που δεν είναι παρόν. Εγώ βεβαίως δεν είμαι ο εκπρόσωπος του, αλλά ούτε και ο κύριος Βαν Ρομπόη παρίστατο τα τελευταία χρόνια σε τέτοιου είδου συζητήσει, γιατί αυτή είναι μια συζήτηση που αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Και αυτή είναι η συμφωνία που έχει συνομολογηθεί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Εξάλλου μην ξεχνάτε, εγώ με τον κύριο Τούσκ έχω συζητήσει διαμακρών τις τελευταίε εβδομάδε. Δεν είναι ότι απλά αυτά που λέμε είναι τυχαία, ε, γιατί αν ήταν έτσι δεν θα είχαμε καταλήξει και στην άποψή μας για την Τουρκία. Η Τουρκία έχει υπετιότητα και η παρουσία του κυρίου Τούσκα στην Τουρκία είναι πολύ πιο σημαντική από το να παρίσταται εδώ στη συζήτηση αυτή ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Και ό,τι και να λέτε έτσι έχουν τα πράγματα. Εγώ λοιπόν έχω προετοιμάσει τη συζήτησή μου αυτή που έλαβε χώρα εδώ με τον πρώτο Συμβουλίου. Ε, ο ίδιος όπως σας είπα έπρεπε να πάει στην Τουρκία και καλώ έκανε. Γι' αυτό την κριτική που ασκήθηκε ει βάρος του την βρίσκω άδικη και παράλογη. Όσον αφορά τώρα στην Ελλάδα. Διότι κάποιοι ε, ανέφεραν αυτό το πρόβλημα. Δεν μιλάμε μόνο για τα 35 δις που προτείνει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξυπακούεται ότι τροφοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Με όλες τις κυβερνήσεις ε, δεν μπόρεσε λόγω διοικητικών προβλημάτων και άλλων να απορροφήσει τα κονδύλια που έχουν τεθεί στη διάθεσή της. Η Ευρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον κύριο Ντομπρόσκι αυτό έκανε. Προσπάθησε να συσσωρεύσει όλου του ανθρώπινους και διοικητικού πόρους που χρειάζονται ούτω ώστε ταχύτατα και με χάρη στου κανόνες συγχρηματοδότηση που διαφέρουν από αυτού που ίσχυαν νωρίτερα για να επιτρέψουν στην Ελλάδα να κάνει αυτό που έπρεπε να έχει ήδη κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και που δεν έκανε ούτε και το έκανε εξάλλου του περασμένου. Ε, μπορώ ώρες να σας μιλάω για την Ελλάδα. Μπορεί κάποιος να ασκήσει ισχυρή κριτική και δεν ε, ισχυρίζομαι ότι από αισθητική ε, πλευρά είναι υπόδειγμα η συμφωνία που διαπραγματευτήκαμε. Αλλά όπως το είχα υποσχεθεί στο Κοινοβούλιο, κάναμε μια αξιολόγηση κοινωνικού αντικτύπου του ελληνικού μνημονίου και εκεί δεν ε, υπήρξε ούτε λέξη επ' αυτού. Εάν είχε υπάρξει, τότε ε, καλά ε, θα κάνατε να μας επικρίνετε επειδή δεν αντικτύπου. Αλλά έγινε. Λοιπόν, για την Ελλάδα, πιστεύετε πραγματικά αν το θέμα του ΦΠΑ και του συντελεστή του για τα, ε, στον τομέα της εστίασης ε, ε, είναι τεχνικό ή πολιτικό ζήτημα. Εμείς παίρνουμε αποφάσεις ως πολιτικοί που είμαστε. Είναι απίστευτο, ίσως δεν το ξέρετε γιατί δεν σας το λένε. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ανέλαβε, ε, ανέλαβε κάτι λογικό να περικόψει το αμυντικό προϋπολογισμό. Αυτό θα έπρεπε να το έχει κάνει η ίδια η κυβέρνηση της Ελλάδας. Ε, και επίσης Υπάρχει το θέμα της δίκαιης φορολόγησης των πλειοκτητών. Δεν το είχε προτείνει η ελληνική κυβέρνηση. Εγώ, χριστιανοδημοκράτης, συντηρητικός, εξεπλάγει διότι ώρες άκουγα μία επιχειρηματολογία από τον Πρωθυπουργό ε, κατά της δίκαιης φορολόγησης των πλουσιωτέρων στην Ελλάδα εις βάρος των φτωχότερων στην Ελλάδα. Δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας που το πρότεινε. Μιλήσατε για ειλικρίνεια. Λοιπόν, ε, δεν είναι σωστό, διότι δεν ακούτε ποτέ και τις δύο πλευράς, ε, πλευρές για, για το ζήτημα. Δεν θέλω όμως να επεκταθώ για αυτό το ζήτημα, διότι θα μου πείτε ότι Μιλάω για εσωτερικά ελληνικά ζητήματα στη σημερινή μας συζήτηση. Όχι, δεν πρόκειται να το κάνω. Πάντως, ε, ο κύριος Τσίπρας ήταν πολύ πιο ευγενικός μαζί μου από ότι εσάς στην τελευταία συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν από λίγες ημέρες. Ναι, η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν μέρος ε, της πρώην Τρόικα, μάλιστα. Εάν δεν υπήρχε όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρόγραμμα προ, προς το μνημόνιο που θα είχε προκύψει θα ήταν κατά πολύ επαχθέστερο σε σχέση με ε, που αυτό που εξασφάλισε η παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ε, ε, διότι από πολλές πλευρές είναι ελαφρύτερο το μνημόνιο σε σχέση με αυτό που θα είχε προκύψει στην αντίθετη περίπτωση. Ας πάρουμε και άλλες χώρες, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Λετωνία. Έδωσαν, απέδειξαν ε, ε, με συγκεκριμένα αποτελέσματα την ανάλυση μου ότι όταν φέρεται σε πέρα στις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις τα προγράμματα είναι πολύ καλύτερα για την ε, συμφωνία TTIP σας άκουσα. Δεν είμαι αφελής. Δεν είμαι αφελή σε ό,τι αφορά αυτή τη συμφωνία ελευθερίου εμπορίου. Απλά αυτό που λένε ότι το χρειαζόμαστε. Τη χρειαζόμαστε τη συμφωνία. Οι όροι με του οποίου θα προκύψει αυτή η συμφωνία είναι θέμα όχι μόνο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και των κρατών μελών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων όσο λαμβάνουν θέση αυτή, ε, χώρα αυτή. Αλλά το να πούμε εκ των προτέρων ότι δεν χρειαζόμαστε μια τέτοια συμφωνία ελευθερίου εμπορίου, όσο και να θέλω δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτή την αντιμετώπιση. Θα πρέπει να κάνουμε σωστέ διαπραγματεύσει, μέχρι τέλου τι διαπραγματεύσει να τι φτάσουμε, αλλά χρειαζόμαστε τη συμφωνία αυτή και θα την πετύχουμε με όρου που ανταποκρίνονται στο ευρωπαϊκό πνεύμα και στι ευρωπαϊκέ ε, αρχέ. Απόλυτα. Για τη Γεωργία τώρα να πάρω το λόγο και να πω δύο λόγια. Δεν μπορούσα να το πω, αλλά Κάποιος ε, το ανέφερε. Εγώ αισθάνομαι πολύ συνδεδεμένος με τους Ευρωπαίους ε, αγρότες. Πάντα και ως πρώην Πρωθυπουργό και υπουργό Οικονομικών προασπίστηκα την ευρωπαϊκή κοινή αγροτική πολιτική γιατί η Ευρώπη χωρίς τους γεωργούς, τους αγρότες, χωρίς ε, αυτούς που φροντίζουν τη γη, τους Τίμωρας δεν θα ήταν η Ευρώπη στην οποία μπορούμε να ζούμε σήμερα. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε ξεκρέμα αυτή τη στιγμή αγρότες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φροντίσει προκειμένου η κρίση στο γαλακτικομικό κλάδο που απειλεί πραγματικά την ίδια την ύπαρξη των επιχειρήσεων αυτών θα φροντίσει να επιληθεί το συντομότερο δυνατόν αυτή η κρίση. Έχουν γίνει κάποιες πρωτοπροτάσεις. Περιμένουμε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τώρα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την μεγάλη προσοχή που αφιέρωσε το Κοινοβούλιο σε μένα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Äh, θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχαριστήσω θερμά κύριε Γιούνκε